Hyvää huomenta. huomenta ja Σας καλημερίζω. Σας εύχομαι επίσης ε, καλή χρονιά. Πράγματι έχουμε σοκαριστεί όλοι από τον αριθμό των θυμάτων στην Αιτή. Μιλάμε πιθανώς για 100.000 νεκρούς. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ας ελπίσουμε ότι οι άνθρωποι η ανθρωπιστική βοήθεια την οποία μπορούμε να παρέχουμε στην ΑΕΤ να λειτουργήσει γρήγορα και αποτελεσματικά και είμαι επίσης βεβαία ότι την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια θα έχουμε την δυνατότητα να επανέλθουμε σε αυτή τη φρικτή καταστροφή και στις συνέπειες που είχε στους ανθρώπους εκεί. Ας επανέλθουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καινούριο. Μπορούμε να την κάνουμε δεκτή. Στις 11.30 διευκρινίζω ότι θα τερματιστεί η συνεδρίαση γιατί μετά θα συνεχιστεί η συνεδρίαση μιας ομάδας εργασίας, μιας ομάδας εργασίας η οποία θα ασχοληθεί με το μέσο δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Θα είναι μια συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να πάρουν μέρος, αλλά μόνο βουλευτές θα είναι η πρώτη επίσημη συνεδρίαση αυτής της ομάδας εργασίας η οποία μόλις πρόσφατα, για την οποία μόλις πρόσφατα είχαμε τις τελικές αποφάσεις για τη σύνθεσή της. Στη συνέχεια κάποιες παρατηρήσεις σχετικά τις ακροάσεις, με τις ακροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων ή των προτινομένων αν θέλετε επιτρόπων. Ε, είμαι βέβαια ότι ακούσατε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή την ακρόαση της Κάθριν Άστον, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ύπατη εκπρόσωπος εξωτερικές υποθέσεις. Έγινε τη Δευτέρα το απόγευμα. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έστειλε μια επιστολή στον Πρόεδρο αμέσως μετά το κλείσιμο της ακρόασης και από πλευράς μας στις 25 ε, Ιανουαρίου μπορούμε να επανέλθουμε στην ακρόαση αυτή για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνεργαστούμε με την ύπατη εκπρόσωπο. Φυσικά ε, στην ουσία θα βασιστούμε στην διοργανική συμφωνία. Δεν θα ζητήσουμε να ανατραπεί οτιδήποτε. Αλλά από την άλλη θα ήταν καλό να μπορέσουμε να γνωστοποιήσουμε τις προσδοκίες μας και τις ελπίδες μας προς την Άστον σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί της. Και θα τη στείλουμε επίσης και μία επιστολή. Περνάμε τώρα στο σημείο 2, ανακοινώσεις της Προεδρίας. Θα προσπαθήσω να είμαι συντομοτέρα της προηγούμενης φοράς, αλλά έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα από την τελευταία μας συνεδρίαση και έτσι δεν μπορώ να τα παραλείψω. Στις 30 Δεκεμβρίου στη Μόσχα προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατέβηκαν σε διαδήλωση. Ανάμεσα σε αυτούς και η κυρία Λουτμίλα Αλεξέγεβα η οποία συνελήφθη αυτή που πήρε το βραβείο Σαχάροφ, συνελήφθη. Δεν ξέρω αν διαβάσατε την International Herald Tribune. Ήταν στην πρώτη σελίδα ε, το θέμα της διαδήλωσης αυτών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία και τις συλλήψεις τους. Θυμίζω ότι υπήρξαν 50 περίπου συλλήψεις μετά από τη διαδήλωση αυτή. μετά από λίγες ώρες κράτησης ε, τους άφησαν ελεύθερους και σχετικά γρήγορα και αυτό συνέβη και για την κυρία Αλεξέγεβα. Γνωρίζετε επίσης ότι ο πρόεδρος μας αντέδρασε σε σχέση με τις συλλήψεις αυτές και απέτησε άμεσα την απελευθέρωσή τους και νομίζω ότι μπορούμε να τον συγχαρούμε γι' αυτό. Πέραν της Ρωσίας, η Κίνα γνωρίζετε ότι την επομένη εβδομάδα θα έχουμε να συζητήσουμε ένα ψήφισμα σχετικό με τον Λιου Τσαου Μπον, έναν διανοούμενο ε, Κινέζου, ο οποίος καταδικάστηκε σε δεκαετή κάθεξη. Γιατί? Γιατί σύμφωνα με τις κινέζικες αρχές ε, είχε ζητήσει, είχε προσπαθήσει να προκαλέσει ε, προβλήματα και είχε παροτρύνει σε εξέγερση του συμπατριώτες του, κάτι το οποίο σύμφωνα με τον Κινέζικο ποινικό κώδικα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Καλό θα είναι να συνεχίσουμε να μην αγνοούμε την υπόθεση του Τσάου Μπον. Ο πρόεδρος Μπούζεκ δημόσια εξέφρασε κριτική για την απόφαση των κινέζικων αρχών. Και να μην ξεχνάμε επίσης και τον Χου Τζα, ο οποίος έχει πάρει το βαβείο Σαχάραφ παλαιότερα. Ο πρόεδρος Μπούζεκ έστειλε μια επιστολή γύρω από την υπόθεση αυτή στον αντιπρόσωπο της Κινέζικης Πρεσβείας της Βεξέλλες. Ας έλθω τώρα σε κάτι το οποίο για μένα στοιχειοθετεί μια καινοτομία. Είναι η κατάσταση των Ουιγούρων, οι οποίοι ε, ε, τους έδιωξαν από την Καμπότζη και αυτή τη στιγμή έχουν σκορπίσει στην Ινδοκίνα. Είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση η κατάσταση των Ουιγούρων. Θυμίζω ότι υπάρχει μια συμφωνία πλαίσιο η οποία συνδέει την Καμπότζη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σε ισχύ από το 2007. Στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής υπάρχει μια ρήτρα η οποία προβλέπει τη διακοπή της συμφωνίας από το 1997 ισχύει η συμφωνία και πρέπει να αντιμετωπίσουμε εκ νέου το θέμα των Ουιγούρων οι οποίοι απελάθηκαν προς την Κίνα. Έρχομαι τώρα στο θέμα του Βιετνάμ. Γνωρίζετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τους μοναχούς και ιερομονάχους οι οποίοι έχουν πέσει θύματα διώξεων στο Βιετνάμ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, παρακολουθεί την κατάσταση και τις τελευταίες εξελίξεις ε, στο Βιετνάμ. Διαπιστώνουμε ότι από το τέλος Δεκεμβρίου δεν έχουν υπάρξει πράξεις βίας εις βάρος ε, της κοινότητας αυτής και η μοναχοί αυτή είναι σε θέση να κηρύττουν το πιστεύω τους ελεύθερα. Ε, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό έχει επηρεάσει η ευρωπαϊκή δράση, όλα αυτά είμαι πεπισμένη ότι είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε τη δράση μας. Ας έλθουμε τώρα στις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας τα διάφορα κατεπήγοντα. Ε, θυμάστε τα κατεπήγοντα τα σχετικά με το Αζερβαϊτζάν και την ελευθερία τύπου. Ξέρετε ήδη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε υπερασπιστεί δύο bloggers οι οποίοι είχαν καταδικαστεί στο Αφγανιστάν. Αυτοί οι δύο ε, εφεσίβαλαν την καταδίκη τους ήδη από τον Δεκέμβριο του προηγούμενου χρόνου. Η απόφαση όμως δεν έχει ληφθεί ακόμα σχετικά με την έφεση και οι δύο αυτοί blogger παραμένουν πάντα στη φυλακή και δεν υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες ε, να ε, υπάρξει αλλαγή στην καταδίκη τους έστω και στη διαδικασία της έφεσης. Εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους απελευθερώσουμε πάρα πολύ σύντομα άλλα δύο θέματα. Πρώτον η Ουγκάντα. Ξέρετε ότι ε, καταλήξαμε σε ένα ψήφισμα το Δεκέμβριο σχετικά με τα σχέδιο νόμου στην Ουγκάντα που προκάλεσε πάρα πολλές αντιρρήσεις εις βάρος των ομοφιλόφιλων. Ζητήσαμε από την κυβέρνηση της Ουγκάντα ο νόμος αυτός να μην γίνει δεκτός γιατί είναι ένας νόμος ο οποίος προκαλεί διακρίσεις εις βάρος των ομοφιλοφίλων μετά από το ψήφισμα αυτό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φαίνεται ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν θετικά. Εν πάση περιπτώσει οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε είναι αντιφατικές και τώρα μου είπαν ότι χθες απεσύρθη το σχέδιο νόμου. Συνεπώς μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι γιατί το ψήφισμα το οποίο υιοθετήσαμε δεν ήταν μάταιο. Πρόκειται για ένα καλό νέο. Κλείνοντας τις ανακοινώσεις θα έλθω στην Δημοκρατία του Κονγκό. Εμείς καταδικάσαμε την βία η οποία έχει ξεσπάσει στην χώρα αυτή, στη Δημοκρατία του Κονγκό Υπάρχει και η Μονίκ, η οποία είναι η αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Εθνών στην Δημοκρατία του Κονγκό και η οποία αποφάσισε να ξεκινήσει μια νέα δράση για να προστατεύσει τους άμαχους πληθυσμούς που πέφτουν θύματα διώξεων και ε, βίας γενικότερα. Είμαι βεβαία ότι θα επανέλθουμε στην κατάσταση στην Ερντεσέ, στη Δημοκρατία του Κονγκό την Άνοιξη, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν συστηματικές μορφές βίας και συστηματική βιασμή εις βάρος των γυναικών. Αυτά είναι τα δραματικά στα οποία είχα να αναφερθώ. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες αντιδράσεις, κάποιος θα ήθελε το λόγο να προσθέσει ένα θέμα δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει το λόγο, πως περνάμε στο σημείο 3. Έχουμε ανάμεσά μας έναν αντιπρόσωπο της Ισπανικής Προεδρίας και ε, θα ασχοληθούμε με το πρόγραμμα της Ισπανικής Προεδρίας για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το λόγο θα δώσω στον Ανδράδε Κουαδράδο είναι διευθυντής ε, του τμήματος ε, ανθρώπινα δικαιώματα στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα συζητήσουμε το θέμα και με τον Νίκολα Μπέλντερ ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για τη διεθνή αμνηστία στην αντιπροσωπεία που έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι η Διεθνής Αμνηστία είναι ένα σημαντικός εταίρος της Επιτροπής μας, της Υποεπιτροπής μας. Ξεκινώντας θα δώσω το λόγο στον κύριο Κουαδράδο. Να τονίσω κύριε Κουαδράδο ότι αναλαμβάνετε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια καθοριστική στιγμή. Το λέω αυτό γιατί πολύ σύντομα περνάμε σε μια νέα περίοδο σχέσεων διεθνών σχέσεων της Ένωσης. Έχουμε ένα πρόεδρο του Συμβουλίου, έχουμε έναν αντιπρόεδρο που, της Επιτροπής που ασχολείται και με τα εξωτερικά θέματα. Βρισκόμαστε σε μεταβατική περίοδο γιατί θα πρέπει να προσαρμοστούμε στο σύστημα αυτό το καινούργιο και περιμένουμε τις απόψεις σας και τις προθέσεις σας για το μέλλον. Κυρίες και κύριοι, μεγάλη μου τιμή που είμαι σήμερα εδώ. Η Ισπανία για τέταρτη φορά μετά την προσχώρηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει την Προεδρία. Αυτή τη φορά όμως η Προεδρία της είναι ιδιάζουσα διότι ακριβώς πέφτει σε μία ουσιαστικότατη στιγμή για την Ισπανία, την Ευρώπη και τη διεθνή συγκυρία. Για την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή και για την Ισπανία το ίδιο. η θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας προσδίδει μια ισχυρή βάση στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Αναλαμβάνει λοιπόν σε μια μεταβατική φάση η Ισπανική Προεδρία το τιμόνι. Είναι τιμή για την τόσο ευρωπαϊκή και ευρωποϊστική χώρα όπως είναι η δικιά μου να παίξει πρωταγωνιστικό χώρο, ε, ρόλο συγγνώμη, στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Αναλαμβάνει όμως την Προεδρία και σε μια φάση ιδιαίτερα κρίσιμη. Κλιματική αλλαγή, ανεργία, οικονομική κρίση είναι οι προκλήσεις της στιγμής και όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία παρεμβαίνουν και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι έξι μήνες λοιπόν που έρχονται είναι σημαντικότατοι για την Ισπανία. και προκλήσεις αλλά και κίνητρα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. Στους επόμενους έξι μήνες και υπό την ηγεσία της Βαρόνης Άστον θα προχωρήσουμε στο σχεδιάγραμμα του πλαισίου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ισπανία δεν θέλει να δημιουργήσει, ούτε και είναι και δουλειά της δηλαδή, να δημιουργήσει μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απλώς θέλει να αξιοποιήσει όλα εκείνα τα μέσα τα οποία ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επεξεργαστεί για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίσει τη συνέχεια στην άσκηση των πολιτικών αυτών. Εμείς δεν θέλουμε να καινοτομήσουμε ούτε να επεκτείνουμε τη γενικότερη πολιτική της Ένωσης. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις ήδη υπάρχουσες πολιτικές και να βγάλουμε από αυτές όλη την προστιθέμενη αξία. Θέλουμε εγκαρσιότητα, συνεκτικότητα και συμβατότητα της πολιτικής της Ένωσης για τα, ευρωπαϊκά, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλουμε διάλογο, διαβούλευση. Διαπραγματεύσεις και με τον ΟΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν θα πρέπει εμείς να μένουμε μόνο σε συνένεση και σε εκπόνηση εγγράφων και σε διακηρύξεις καλών προθέσεων. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε σαφείς γραμμές στα κράτη-μέλη στις πρεσβείες μας για, την προστασία όλων όσων παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα συνεχίσουμε την πολιτική της Σουηδικής Προεδρίας για την υλοποίηση των κατευθυντηρίων γραμμών. Θα προσέξουμε ιδιαίτερα και τα τις προσωπικές περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και με την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε συνένεση μεταξύ των 27. Θα συνεργαστούμε στενά και με την Κομισιόν και τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και με τη Βαρόνη Άστον φυσικά. Θα έχουμε συνεχή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνοντας υπόψη όλες τις δράσεις του Κοινοβουλίου, ενημερώνοντας το Κοινοβούλιο τι γίνεται και στην Ειδική Επιτροπή, στο ΚΟΜ και θα ζητήσουμε από την κυρία Χάουταλα να συμμετέχει στο ΚΟΜ άμεσα και να ενημερώνεται επίσης άμεσα για το περιεχόμενο όλων των συζητήσεων. Θα πρέπει επίσης να συνεργαζόμαστε στενά με τις αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πρεσβείες μας όπως επίσης και τις αντιπροσωπείες μας στους διεθνείς οργανισμούς. Παλεύοντας για τη διάδοση όλων εκείνων των αρχών που εμπνέουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ανά τον κόσμο. Μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι αγώνας κατά της θανατικής ποινής, αγώνας κατά των βασανιστήριων, προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, προστατε... απαγορεύοντας ε, καταπολεμώντας μάλλον το φαινόμενο των παιδιών στρατιωτών καταπολεμώντας την ομοφοβία δικαίωμα στο νερό προστασία των αναπήρων προστασία των αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, θέλουμε να ενισχύσουμε τον ΟΗΕ και τον οργανισμό που θα δημιουργήσει το 2011 για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λοιπόν, τώρα για το εξάμεινο. Ο Σαπατέρο θεωρεί προσωπική του υπόθεση την καταπολέμηση της θανατικής ποινής. και στις διμερείς επαφές που είχαν κυβερνητικοί παράγοντες της Ισπανίας με τρίτες χώρες η κατάργηση της θανατικής ποινής ήταν ένας από τους βασικούς άξονες. Και αυτό θα γίνει και μία προτεραιότητα για την Προεδρία μας κατάργηση της θανατικής ποινής στις αραβικές χώρες. Είχαμε τη δήλωση της Μαδρίτης σχετικά. Και ο, κύριος Σαπατέρο ξεκίνησε και μία διεθνή επιτροπή καταπολέμηση της θανατικής ποινής κατάργηση της θανατικής ποινής και την πρόθεση του διαλόγου για την κατάργησή της. Για να λειτουργήσει γρήγορα και εύρυθμα αυτή η Επιτροπή διορίσαμε έναν εθνικό συντονιστή για την κατάργηση της θανατικής ποινής στο βαθμό του πρεσβευτή, του πρεσβευτή Α. Ο Ραφαέλ Βάγε είναι σήμερα αυτός ο πρεσβευτής και θα αποτελέσει και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μελλοντικής Επιτροπής του ΟΗΕ. Η Ισπανία λοιπόν θα συνεχίσει να παλεύει στους άξονες που ήδη έχει προχαράξει για την κατάργηση της θανατικής ποινής. Η Βαρόνι Άστον και ο Άγχελ Μορατίνος συναντήθηκαν τον προηγούμενο μήνα στη Μαδρίτη και συζήτησαν το θέμα. και στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους διεθνείς οργανισμούς αποφασίστηκε να προσληφθούν εμπειρογνώμονες σε ποινικά ζητήματα. Όπως επίσης ανάληψη από Ευρωπαίους αρμόδιους ή προστασία των Ευρωπαίων πολιτών που καταδικάζονται σε θάνατο σε τρίτες χώρες. Οι διμερείς επαφές των κρατών μελών θα πρέπει να γίνονται παράλληλα και συντονισμένα με αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να προχωρήσουμε για το 62, 149 και 63, 153 τα δύο ψηφίσματα και το μορατόριου του ΟΗΕ για τη θανατική ποινή. Το 2010 λοιπόν θα είναι μια ουσιαστικότατη χρονιά. Θα πρέπει να παλέψει ούτως ώστε να υπάρξει συσπήρωση γύρω από αυτό το ψήφισμα. Και με το Βέλιο εμείς προχωρούμε συντονισμένα στην διατύπωση του νέου ψηφίσματος. Και στο ΚΟΜ ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα η συζήτηση μεταξύ των 27. Εμείς θα συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την καταστρεπτική δράση αυτών που αντιτίθενται στην κατάργηση της θανατικής ποινής για να εξαφανιστεί η θανατική ποινή από τον κόσμο. Θέλουμε άμεσα να καταργηθεί η θανατική ποινή σε καταδικασμένους ψυχοπαθείς ή καταδικασμένους που ήταν ανήλικοι όταν εγκλημάτισαν και έγκες γυναίκες. Θέλουμε λοιπόν να περάσουμε αυτό το θέμα εγκάρσια σε όλες τις διαβουλεύσεις και συζητήσεις και διαπραγματεύσεις που θα έχουμε στο μέλλον. Επίσης, θέλουμε να εγκρίθει και η Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα Θέλουμε να παρέμβουμε και στις καταδίκες εκείνες για πολιτικούς λόγους. «24 με 26 Φεβρουαρίου θα έχουμε το τέταρτο παγκόσμιο συνέδριο κατά της θανατικής ποινής. Και αυτό το γεγονός εμείς το θε, βάλαμε στην ημερήσια διάταξη της ΚΟΜ ούτως ώστε να συμμετέχουν σε είπα, το επίπεδο οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στις τρίτες χώρες. Στην περίπτωση της Ισπανίας εμείς θα εκπροσωπηθούμε από τον Πρωθυπουργό μας τον Σαπατέρο τα βασανιστήρια παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε όλα τις επίπεδα και λίγες είναι οι χώρες που μπορούν να πούν ότι δεν ασκούνε βασανισμό. Γι' αυτό λοιπόν η καταπολέμηση αυτής της μάστιγας αποτελεί προτεραιότητα της Ένωσης εδώ και χρόνια. Να καταπολεμήσουμε λοιπόν τα βασανιστήρια, τις συμπεριφορές εκείνες που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όπως επίσης όμως θα καταπολεμήσουμε και την τρομοκρατία. Θα παρακολουθήσουμε από κοντά και τις προσωπικές περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με διαβουλεύσεις, θα συνεργαστούμε με την Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των βασανιστήριων, και με τις αντίστοιχες επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων οργανισμών. Η Ισπανία επικύρωσε ήδη το προαιρετικό πρωτόκολλο κατά των βασανιστήριων. Και μέσω του διαμεσολαβητή η Ισπανία ήδη έχει αναθέσει την εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλου σε ισχύ για την πρόληψη των βασανιστήριων. Η Ισπανία είναι είναι υπέρ του διορισμού της κυρίας Άντος Ρούης ως αρμόδιας για την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών. Αυτή η ειδική αντιπρόσωπος θα υποστηριχθεί από την Οσπανική Προεδρία με όλα τα μέσα. Εμείς θα προωθήσουμε συντονισμένη εργασία στις 10 χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το ειδικό πρόγραμμα του Οργανισμού για την Προστασία των Παιδιών και θα παλέψουμε για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών όπου αυτά τα δικαιώματα παραβιάζονται είτε με, καταναγκαστική εργασία, είτε με βία, είτε με οτιδήποτε άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να εξετάσει το πρόβλημα των παιδιών στρατιωτών. Είναι τα παιδιά τα οποία είναι στρατιώτες σε εμπόλεμες περιοχές. Θέλουμε να δούμε επίσης και τι γίνεται με την διαφορά φύλου στην περίπτωση των παιδιών στρατιωτών. Διότι τα κοριτσάκια στρατιώτες είναι ιδιαίτερα πιο ευπαθή. μέσα στο γενικότερο πρόβλημα. Δήλωσε λοιπόν ο πρόεδρος μας, ο πρωθυπουργός μας, συγγνώμη, ότι θα το επόμενο εξάμεινο θα σφραγιστεί η Προεδρία μας από την καινοτομία για την προστασία και πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. η ευρώπη θα προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φίλων, μεταξύ των κρατών μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων. θα παλέψουμε για την η ισότητα ανδρών γυναικών για την καταπολέμηση των σεξουαλικών διακρίσεων. σε όλα τα φόρα και σε όλες μας τις πολυμερεί διαπραγμα... Ε, διαπραγματεύσεις και διεθνείς οργανισμούς. Η Μαρία Τερέζα Φερνάντε Δελαβέγα, πρώτη αντιπρόεδρο τη Ισπανική κυβέρνηση, το έχει πραγματικά στην καρδιά τη αυτό το θέμα των σεξουαλικών διακρίσεων και έχει φτιάξει και μία ειδική γενική γραμματεία. Θέλει να προασπιστεί η ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα, στην πολιτική, στην κοινωνία, στην εργασία και στην Βαλένσια θα γίνει τον επόμενο μήνα μία συνάντηση για αυτά τα θέματα. Εσείς λέτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά μιλάτε πάρα πολύ γρήγορα. Υπό την Προεδρία έλεγα της αντιπροέδρου της κυβέρνησης θα γίνει στη Βαλένθια η συνδιάσκεψη για τις γυναίκες σε έναν καλύτερο κόσμο. Οι προηγούμενες συναντήσεις είχαν ως σκοπό την ανταλλαγή εμπειρίες μεταξύ Αφρικανών και Ευρωπαίων γυναικών. Τώρα θα διευρύνουμε εμείς τη συμμετοχή και με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Θα ενισχύσουμε λοιπόν όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτής της νέας Ευρώπης. Στα πλαίσια της ΚΕΠΑ η η ισότητα των φύλων αποτελεί ένα εγκάρσιο αίτημα σε όλες μας τις διαπραγματεύσεις και συναλλαγές. Αποτελεί μάστιγα η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, όπως και οι άλλες μορφές διακρίσεων. με την τσεχική και σουηδική προεδρία οι πρεσβείες των 27 προχώρησαν σε επιτόπου αναλύσεις της κατάστασης και η Task Force που εξετάζει τα προβλήματα βίας κατά των γυναικών της ΚΟΜ εξετάζει αυτά τα στοιχεία που αποτελούν πλέον μια πηγή δεδομένων και θέλουμε να προχωρήσουμε πιο μακριά. Να έχουμε δηλαδή σαφείς δεσμεύσεις και πρακτικά αποτελέσματα και στην Ευρώπη τα οποία θα προωθήσουν οι πρεσβείες μας ανά τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κοιτάξει τη διαμόρφωση τοπικών στρατηγικών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Η Προεδρία θα εξετάσει από κοντά και προσωπικές περιπτώσεις γυναικών που των οποίων παραβιάζονται τα δικαιώματα ή που υπόκεινται βία. Ας πούμε, ε, αγωνίστριες ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θα δούμε επίσης την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες και όλα αυτά θα συμπεριλαμβάνονται σε όλον τον τύπο της, ως όλων των τύπων της επαφές. Η Ισπανική λοιπόν Προεδρία θέλει να εξετάσει πώς εφαρμόζονται στην πράξη πώς εφαρμόζονται στην πράξη πώς εφαρμόζονται στην πράξη τα ψηφίσματα του ΟΗΕ 13, 25, 18, 20, 18, 89. Και όλα αυτά γίνονται όλα αυτά πέφτουν σε μια καταπληκτική συγκυρία διότι έχουμε τα 15 χρόνια της επαιτίου της διάσκεψης του Πιτζίν και από 1η μέχρι 12 Φεβρουαρίου θα γίνει στη Νέα Υόρκη η τέταρτη συνδιάσκεψη του CSW. Προτεραιότητα λοιπόν της Ένωσης στη διάσκεψη της CSW είναι να συνεχιστούν, να προχωρήσουν μάλλον οι αποφάσεις της διάσκεψης του Πεκίνου. Τώρα, σεξουαλικές επιλογές και προσανατολισμοί επίσης θα πρέπει να διασφαλιστούν. Διότι σε ορισμένε χώρες ε, άτομα τα οποία έχουν διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις από ότι οι ισχύουσες ε, στην κοινωνία τους υπόκεινται διακρίσεις, διώξεις, βασανισμούς και πολλές φορές αδιάκριτα δολοφονούνται. Σε πολλές χώρες συνενετικές σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ενηλίκων καταδικάζονται από, τον ποινικό, ε, ε, ε, από τα δικαστήρια. Δηλαδή, οι λεσβίες, γκέι, και λοιπά διώκονται. χωρίς να υπερβάλλουμε τα τελευταία χρόνια η Ισπανία είναι πιονέρος στην προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Έχουμε ελευθερία στο γάμο των ομοφιλοφίλων, ε, επιτρέπεται οι ομοφιλόφιλοι να υιοθετούν παιδιά. Και θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις σε χώρες όπως στο Ιράκ και σε άλλες χώρες, αραβικές χώρες. Πολλές φορές λοιπόν βλέπουμε ε, ότι ενώ έχουμε δυνατότητες να υπερασπιστούμε εμείς τους LGBT, lesbian, gay, trans, ε, ενώ έχουμε λοιπόν τα μέσα στη διάθεσή μας νομικά να το κάνουμε, δεν προχωρούμε στην πράξη. Θέλουμε λοιπόν το κόμμα να εγκρίνει ένα toolkit ένα κουτί εργαλεία δηλαδή που θα μπορεί να χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθάει τους LGBT ανά τον κόσμο. Πράγμα το οποίο ήδη κάνουν η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία και η Σουηδία. Η Προεδρία λοιπόν θα συγκαλέσει μία τουλάχιστον συνεδρίαση της συμβουλευτική Επιτροπής ε, για τον LGBT στα πλαίσια του κόμμου. όπου θα συμμετέχουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. 67 χώρες υπέγραψαν το ψήφισμα για την αποποινικοποίηση της ομοφιλοφιλίας ανά τον κόσμο. Και έχουμε συντονίσει με το Βέλγιο που θα διασφαλίσει την επόμενη Προεδρία την δράση μας ούτως ώστε να παραμείνει ζωντανή η όθηση του, της δήλωσης του 2008. Μεγαλύτερη ρώση λοιπόν συντονισμό μεταξύ της ΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ του Συμβουλίου της Ευρώπης και των άλλων οργάνων που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η κυρία Πιλάγιο που είναι η πατιαρμοστής έχει δεσμευτεί σχετικά. Τώρα με τους ε, transsexual, τι γίνεται. Οι γκέι και οι λεσβίες Οι διακρίσεις λοιπόν των φιλομεταβατικών είναι διαφορετικές από ότι των γκέι και των λεσβιών. Θα οργανωθεί λοιπόν στη Βαρκελόνη η πρώτη διεθνής διάσκεψη για τα δικαιώματα των φιλομεταβατικών. Λοιπόν, πρόσβαση στο πόσιμο νερό. Τα τελευταία χρόνια είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται ιδιαίτερα στον ΟΗΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν παρούσα σε, όλα, σε όλες αυτές τις δράσεις. Θέλει λοιπόν να αλλάξει εντελώ πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, να αντιστρέψει τα πράγματα και να γίνει προ... Ε, πιονέρος στην πρόθεση αυτού του δικαιώματος. και θα συνεχιστεί, θα δοθεί μια ευρωπαϊκή υπόσταση στην πολιτική που έχουν αναλάβει ήδη η Ισπανία και η Γερμανία στα πλαίσια του ΟΗΕ. και η κυρία Αλμπουκέρκε θα συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαμόρφωση μιας διαπεριφερειακής στρατηγικής. για να μπορέσουμε δηλαδή με αυτές τις θέσεις να πάμε στην 215η συνδιάσκεψη για το νερό το Σεπτέμβριο του 2010. Προστασία των αναπήρων. Άλλη προτεραιότητα. Η Ισπανία υποστήριξε την Τσεχική και Σουηδική Προεδρία για να καταλήξουμε στην προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση του ΟΗΕ για την προστασία των δικαιωμάτων των αναπήρων. Όλα, όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις βέβαια είχαν, ευόδωσαν αλλά έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Θέλουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στην πρώτη σύμβαση του αιώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στους επόμενους έξι μήνες θα προωθήσουμε την επικύρωση της σύμβασης από τις χώρες που δεν το κάναν ακόμα και θα υποβάλουμε στην ομάδα εργασίας του ΚΟΟΜ έναν κώδικα συμπεριφοράς για τους 27 και τα ευρωπαϊκά όργανα. Όπως είπα και στην αρχή, καμία από τις προτεραιότητες δεν θα επιτευχθεί άμα δεν προστατεύσουμε τους αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες. Θέλουμε να διαδώσουμε την θέση μας για την προστασία των αγωνιστών και αγωνιστρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την διαμόρφωση τοπικών στρατηγικών θέλουμε να εμπλέξουμε όλους αυτούς τους αγωνιστές στην ίδια την προστασία, την, στην αυτοπροστασία τους. Θα προχωρήσουμε λοιπόν σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση των υπαρχουσών στρατηγικών, θα επεξεργαστούμε κάποιες μερικές καινούργιες και θα προχωρήσουμε σε συνεδριάσεις επιτόπου όπου θα συμμετέχουν αντιπροσωπείες και πρεσβείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης και τοπικές αρχές Θέλουμε να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών που θα βελτιώνει τις σχέσεις μεταξύ Ένωσης και αγωνιστών. Τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί οι διάλογοι και διαβουλεύσεις με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και συντονίζονται όλα αυτά από την ομάδα εργασίας ΚΟΜ. Δεν έχουμε εδώ το χρόνο για να αναλύσουμε εδώ την κάθε διαβούλευση, διάλογο ή στρογγυλό τραπέζι που θα έχουμε στο μέλλον. Η Σίλβια Εσκομπάρη, η συνάδελφός μου που το παρακολουθεί μερικά από αυτά, θα έρθει να σας τα πει μια άλλη φορά. Πολύ γρήγορα. Να αναφέρω διαβουλεύσεις με τη Ρωσία, την Κίνα, την Αφρικανική Ένωση. Κεντρική Ασία. με τη Ιαπωνία, με την Αμερική, με τον Καναδά και τις υποψήφιες χώρες ε, έχουμε θεσπίσει διάλογο και θα έχουμε διάλογο και με την Ινδονησία στην Τζακάρτα στο εγγύς μέλλον. Και θα έχουμε και τον πρώτο γύρο με τη Μολδαβία. Να πω επίσης και ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διεθνείς οργανισμούς. Θα έχουμε τη 13η και 14η συνεδρίαση της Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στα πλαίσια του ΟΗΕ και εμείς εκεί θα προσπαθήσουμε προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και να, να ενισχύσουμε τη θέση της αρμοστού για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυξάνονται συνεχώς οι επίσημες και ανεπίσημες συναντήσεις στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι απόλυτα ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν θα αντιπροσωπεύεται στα διεθνή όργανα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα χρησιμοποιήσουμε ό,τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας για να ορίσουμε μια κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και μια στρατηγική κοινή για να μπορούμε να έχουμε εξωτερικές και εξωτερική υποστήριξη. Αυτό θα εξαρτηθεί από την ικανότητα που έχουμε να ετοιμαστούμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να προστοτεύουμε την ανεξαρτησία του γραφείου της ΥΠΑ της Αρμοστού του ΟΗΕ και την ανεξαρτησία κάθε διαλόγου και διαπραγμάτευσης. Και επειδή μίλησα πολλή ώρα, επαναλαμβάνω ότι είμαι στη διάθεση της Επιτροπής σας και επαναλαμβάνω και την πρόσκλησή μου στην κυρία Χάουταλα να συμμετέχει στις συνεδριάσεις μας. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, παρουσία σας αυτή. Εάν δεν ήταν σημαντικά τα όσα είχατε να παρουσιάσετε θα σας είχα διακόψει, αλλά αφού είναι τόσο πράγματι φιλόδοξο το πρόγραμμα της Προεδρίας σας, δεν ήθελα να το κάνω. Θα ήθελα λοιπόν να σας συγχαρώ για την ανάληψη της ε, Προεδρίας από την Ισπανία και ελπίζουμε πως ε, θα είναι υποδεγματική σε ό,τι αφορά δηλαδή και την συνοχή μεταξύ της ε, πολιτικής ε, της Προεδρίας και το είπα του εκπροσώπου. Ε, να δώσω όμως καταρχήν το λόγο στον David Nichols από τη Διεθνή Αμνηστία. Είναι σωστό το όνομα που έχω. Μήπως έκανα λάθος. Ναι, θα ήθελα να στήσω συγγνώμη εκ μέρους του Νικολάς, γιατί πράγματι δεν είμαι εγώ αυτός, δεν, δεν μπορούσα να παρευρεθεί σήμερα εδώ. Ε, όπως ε, ήδη ανέφερε η Ισπανική Προεδρία αναλαμβάνει σε μια περίοδο ιδιαίτερης αβεβαιότητας ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας της εξωτερικής ε, πολιτικής. Ε, τόσο κατά την Ισπανική όσο και κατά την Βελγική Προεδρία εγώ θα συμμετέχω στην εφαρμογή και στο σχεδιασμό αυτού του νέου συστήματο. Εκείνο που είναι λοιπόν κέρια σημασία σε αυτή την αβέβαια περίοδο είναι να μην δημιουργηθεί ένα κενό, αν θέλετε, ε, ηγεσία, α το πούμε έτσι, δηλαδή τελικά να βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου κανείς δεν θα ξέρει ποιο είναι υπεύθυνο γιατί και ποιο κάνει τι. Να μην υπάρχει δηλαδή ανάληψη τη ευθύνη για το τι συμβαίνει. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό σε ό,τι αφορά τι δράσει που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή τόσο στη Γενέβη όσο και στην Νέα Υόρκη. Αλλά ε, και οι δράσει που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των αντιπροσωπιών τη στι διάφορε πρωτεύουσε. Γίνονται λοιπόν ε, κάποιε αλλαγέ ε, σταδιακά και θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο με τα τρίτα μέρη και τις τρίτες χώρες το ποιο είναι υπεύθυνο για την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανα πάσα στιγμή. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα ακόμα γενικό σχόλιο πρωτού αναφερθώ στα όσα παρουσίασε η Ισπανική Προεδρία ως πρόγραμμα της. Να πω λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της Ουδικής ε, Προεδρίας είδαμε κάποιες πολύ θετικέ ε, πρωτοβουλίες ε, και υπήρξε, πραγματικά έγινε, ήταν πολύ επιτυχή σε ό,τι αφορά την διαφάνεια. Ε, όμως δεν βλέπουμε να συνεχίζεται αυτή η πρακτική τώρα σε αυτή την Προεδρία. δεν ξέρουμε κατά πόσο βέβαια αυτό οφείλεται στα διοργανικού χαρακτήρα ζητήματα που εξακολουθούν να εκκρεμούν ή εάν υπάρχουν κάποια προβλήματα ε, με την Προεδρία ως προς τον τρόπο που λειτουργεί στο σελίδα της και ούτω καθεξής. Ε, θα ήθελα, εν πάση περιπτώσει, να τονίσω για μία ακόμα φορά ε, τη σημασία, το ρόλο της διαφάνειας σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες της Προεδρίας, όπως αυτή είχε, σας λέω, θεσπιστεί από τη Σουηδική Προεδρία ε, σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα δηλαδή στα δεδομένα από την πλευρά της Προεδρίας. Η Σουηδία πάντα τέτοιου είδους πληροφορίες είχε διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της και τις διέθετε στο ευρύτημα μπορεί να φαίνεται πω αποτελεί μια λεπτομέρεια, αλλά πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο στι εργασίε όλων των οργανώσεων τη κοινωνία ε, των πολιτών, αλλά και για όλου. Ε, και, νομίζω και, και στι εργασίε των ίδιων των Ευρωβουλευτών, ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή την προετοιμασία και των συναντήσεων των ομάδων του Συμβουλίου. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρόγραμμα εργασία που μόλι τώρα μα παρουσίασε η Ισπανική Προεδρία. Ε, ίσως ε, θα είδατε ένα ε, έγγραφο συστάσεων το οποίο αποστήλαμε εμείς στη Σημανική Προεδρία το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ έξω από την αίθουσα αλλά είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα μας. Ε, χωρίς να θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες θα ήθελα να α, πω ότι έχουμε συμπεριλάβει 10 διαφορετικές περιπτώσεις στο, α, στο τέλος εδώ του φυλαδίου για τα οποία 10 ζητήματα απαιτούμε να αναλυθεί συγκεκριμένη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώ και θέλουμε να ε, αναλυθεί δράση σε περισσότερα θέματα, αλλά μιλάμε για 10 συγκεκριμένα σημεία τα οποία είναι η γενικότερου εύρου, αν θέλετε, και πολιτικού βάρου. Γνωρίζω πως ε, υπήρξε στο παρελθόν ε, πρόβλημα σε ό,τι αφορά το, το να θίγονται συγκεκριμένε ε, περιπτώσει και συγκεκριμένα κράτη-μέλη, αλλά νομίζω πω τώρα, μετά, στην περίοδο μετά από τη Λισαβόνα, θα πρέπει να επιληθεί αυτό το ζήτημα. Θα θέλαμε λοιπόν να λάβουμε την ε, βοήθειά σα σε ό,τι αφορά την επίλυση αυτών των 10 συγκεκριμένων ζητημάτων ή προβλημάτων που θέτουμε προ τη Ισπανική Προεδρία. Σε ό,τι αφορά τώρα του ε, τους τομείς της προτεραιότητας στους ανέφερε η Ισπανική Προεδρία. Ε, προφανώς πρόκειται για κοινού ε, στόχου μεταξύ δηλαδή τη Προεδρία και της Αμνηστία και άλλων διεθνών οργανώσεων. Ε, μας χαροποιεί το γεγονός ότι αναφέρατε την, ε, τον αγώνα για την κατάργηση της ανατικής καταδίκη. Ε, γιατί πράγματι θεωρούμε και εμείς ε, πως είναι πολύ σημαντικό, ειδικότερα ε, καθώς κινούμαστε προς τη σχετική ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ στα τέλη αυτού του έτους θα πρέπει να μάθουμε όλοι τα μαθήματα μας από το 2007 και το 2008 σε σχέση με τη συνεργασία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες ε, περιοχές του κόσμου και τον ρόλο που έβεξαν οι οργανώσεις της ε, κοινωνίας των πολιτών σε αυτές τις επαφές. Επίσης θα θέλαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναμειχθεί περισσότερο σε αυτή τη διαδικασία και ειδικότερα τα μέλη του τα οποία ε, ενδιαφέρονται ε, για αυτέ τι προσπάθειε για την κατάρριξη τη θανατική ε, καταδίκη να έρθουν σε επαφή μαζί μα και ε, σε συντονισμό με την Ισπανική Προεδρία να δούμε πώ μπορούμε να εργαστούμε περαιτέρω σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα επίση αυτή την πρόσκληση να την επεκτείνω σε ό,τι αφορά τη γενική διάσκεψη που θα λάβει η χώρα στα τέλη Φεβρουαρίου στη Γενέβη που έχει το ίδιο θέμα, δηλαδή την κατάσταση καταδίκηση. Μετά ε, η αναθεώρηση ε, ε, που θα γίνει σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο του, των Ηνωμένων Εθνών γνωρίζουμε πως είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τη δική σας πλευρά και ελπίζουμε πως οι ευρωβουλευτές θα αναμειχθούν στις διαδικασίες επαφών με άλλες χώρες που είναι οπωσδήποτε απαραίτητες ειδικότερα όταν θα γίνει και η σχετική ε, συνάντηση το Μάρτιο. Επίσης, εκείνο που θα είναι κέρια σημασίας είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έκθεση Goldstein. Ε, το ζήτημα αυτό αποτέλεσε στο παρελθόν ε, ιδιαίτερο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζουμε πως η Γενική Συνέλευση όσο και το συνεδρίο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Ονομάτων το Μάρτιο, δεν έχουν προβεί σε στάσεις και δύο πλευρές σε ό,τι αφορά την διαξαγωγή συγκεκριμένων ε, ερευνών. Αλλά μόνο με βάση ε, τέτοιες συγκεκριμένες και ενδελεχείς ερευνές ε, μπορεί να δοθεί μια σωστή απάντηση στι δύο αυτέ συνεδριάσει, δηλαδή Γενική Συνέλευση και Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, τι εργασίε που γίνονται σε σχέση με τα βασανιστήρια, μα χαροποιεί ε, αυτό που είπε η Ισπανική Προεδρία, ότι δηλαδή θέλει εδώ να συνεχίσει τι προσπάθειε και να συνεχίσει γιατί τα όσα ξεκίνησε η Σουδική Προεδρία σε ό,τι αφορά τι ε, κατευθυντήριε γραμμέ ε, για τα βασανιστήρια. Ε, γνωρίζετε αυτέ οι κατευθυντήρε γραμμέ είναι συγκαταλέγονται σε οι οποίε δεν έχουν εφαρμοστεί ε, ιδιαίτερα σωστά και όπως ε, ε, γνωρίζετε η Σουηδική Προεδρία έχει ξεκινήσει μια σχετική πρωτοβουλία την οποία ελπίζουμε πως θα συνεχίσετε από την πλευρά της δικής σας Ισπανικής Προεδρίας. Σε ό,τι αφορά τα βασανιστήρια, εκεί που θα θέλαμε να λάβουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ε, μια αναθεώρηση του σχετικού ε, κανονισμού ε, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το εμπόριο των εργαλείων βασανιστήριων. Γνωρίζουμε δηλαδή πως αυτός ο κανονισμός δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί πλήρως σε όλα τα κράτη-μέλη και υπάρχουν και κάποια κενά μέσα σε αυτό το κανονισμό τα οποία επιτρέπουν ε, στο, στα κράτη-μέλη να καταστρατηγήσουν τις διατάξεις και δηλαδή να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας ε, αυτών των εμπορευμάτων. Ε, θα ήθελα να θέξω ένα-δύο ζητήματα που έθεσε η Ισπανική Προεδρία σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας και το θέμα της διεύρυνσης. Όπως γνωρίζετε, Ε, κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας θέλουμε να εξετάσουμε ε, διάφορες ε, συμφωνίες σύνδεσης οι οποίες βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, κυρώνονται, υπογράφονται και ούτω καθεξής και βέβαια το, τα σχετικά σχέδια δράσης. Σε σχέση λοιπόν με όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχει εδώ μία ευκαιρία που έχουμε να διαμορφώσουμε την πολιτική γειτονία που εφαρμόζουμε ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα ε, δικαιώματα. Και εδώ αναφέρομαι ειδικότερα στην περίπτωση του Μαρόκου καθώς θα μπορούσε να ε, ε, αποτελέσει ένα υπόδειγμα για όλες τις συμφωνίε σύνδεση που ενδεχομένω θα ακολουθήσουμε βορειοαφρικανικές χώρες. Επίσης θα θέλαμε να βλέπουμε να αναβιώνεται ε, η Συμφωνία της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας ε, και να δούμε πιο ακριβώς ε, εδώ είναι το σχέδιο δράσης. Και επιτρέψτε μου επίσης να πω κάτι πολύ σύντομα σε ό,τι αφορά τις αλλαγές που έγιναν στην περίοδο μετά τη Λισαβόνα και το πώς εμείς φανταζόμαστε ότι τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται στις έρευνες εξωτερικών δράσεων. Είναι θετικό το γεγονός ότι θα υπάρχει ε, μία επαφή μεταξύ αυτής της ομάδας και της Επιτρόπου Άστον. Και εδώ θα σας παραπέμψω σε μια επιστολή που της είχαμε αποστείλει πριν από τα Χριστούγεννα ως προς το πώς μπορούν να ενταχθούν στις βασικές πολιτικές της Ένωσης ε, ε, τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εδώ θα αναφέρω δύο συγκεκριμένα σημεία. για παράδειγμα, οι διαγραφικέ ομάδε εργασία αλλά και οι ομάδε υψηλού επίπεδου του Συμβουλίου, δηλαδή η Κορεπέρ, ε, αλλά και το ε, Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων αποτέλεσαν όλα τους φορά όπου ήταν δύσκολο να ενταχθούν μέσα στις βασικές πολιτικές τους τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα θα θέλαμε λοιπόν ε, η η Επίτροπος Άστον αποφασίσει να υπάρχει ένα μόνιμο ε, πρόεδρο ε, στο Ισοτικό ε, Συμβούλιο για να ώστε να διασφαλίσει ότι ακριβώ θα υπάρχει αυτό ο παράγοντα, αυτή η παράμετρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, επίσης θα θέλαμε να αναλυφθεί μεγαλύτερη ευθύνη σε ό,τι αφορά τη σχετική πολιτική και μεγαλύτερη ευθύνη και από την πλευρά των αντιπροσωπιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των σχετικών κατευθυντήρων γραμμών. Ε, προφανώς εδώ θα κληθούν ε, ένα μέρος αυτών των εργασιών να ε, επιτελέσουν οι πρεσβείες των διαφορών κρατών μελών στις ενλόγων χώρες, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ένα σημείο επαφής στις αντιπροσωπείες ούτως ώστε να υπάρχει μια δυνατότητα διαβίβασης πληροφοριών προς τον υπατό σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Επιστήσατε την προσοχή μας και στην επιστολή την οποία έχετε αποστείλει στην ύπατη εκπρόσωπο σχετικά με τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό το βρίσκω θετικό. Είναι αλήθεια ότι πάρα πολύ σύντομα και εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστούμε με την κυρία Άστον και γι' αυτό η επιστολή σας θα είναι χρήσιμη αλλά κάθε πράγμα στον καιρό του. Και τώρα θα δώσω πλέον το λόγο στους ανυπόμονους πια συναδέλφους. Ξέρετε ότι έχουμε και να συζητήσουμε μετά τη Συρίας, όπως επίσης και το κεκλεισμένο των θυρών μετά τις 11 και μισή και γι' αυτό σας ζητώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι όλοι. Ακούσαμε με πάρα πολύ προσοχή και λεπτομερέστατα τους στόχους της Ισπανικής Προεδρίας και της Amnesty International. Γι' αυτό λοιπόν η κυρία Χιμένες έχει το λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν κυρία Κουαδράδο και να σας ευχαριστήσω και για την παρουσία σας εδώ σαν εκπροσώπου της Ισπανικής Προεδρίας. Αναφέρθηκε ο κύριος ε, Ντουάρτε και στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ομάδων των πολιτών που έχουν ανάγκη από την υπεράσπιση αυτή των πιο ευάλωτων ομάδων και δεν μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε ε, αυτά τα προγράμματα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη από την υποστήριξη αυτή. Δυστυχώς η δική μου χώρα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στον χώρο της τρομοκρατίας που έχει φρικτές συνέπειες για τους αθώους μερικές φορές πολίτες. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να βρίσκουμε τρόπους καταπολέμησης της τρομοκρατίας και να υπερασπιζόμεθα τα δικαιώματα των θυμάτων της τρομοκρατίας. Έχω συζητήσει το θέμα ήδη με την κυρία Μέλστρομ να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια χάρτα δικαιωμάτων των θυμάτων της τρομοκρατίας, των τρομοκρατικών ενεργειών. Όλοι είμαστε υποψήφια θύματα τέτοιων ενεργειών και έχουμε κάθε δικαίωμα να αποκαθίσταται η δικαιοσύνη και να προασπιστούν τα δικαιώματά μας. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τι σκοπεύει να κάνει προς την κατεύθυνση αυτή η Ισπανική Προεδρία. Θα ήθελα επίσης να πω ότι ο συνάδελφος Γιάννης, ο Λουίς Γιάννης, ξέρετε ότι στις αρχές του μηνός Ιανουαρίου μετέβη στην Κούβα με τη σύζυγό του. Σας ζητώ να κλείσετε παρακαλώ, δεν έχουμε χρόνο. Τι σκοπεύει να κάνει η Ισπανική Προεδρία γύρω από την υπόθεση αυτή. Ξέρετε ότι συνελήφθη και απελάθη. Βλέπουμε λοιπόν την περίπτωση ενός Ευρωβουλευτή ο οποίος δεν μπόρεσε να εισέλθει στην Κούβα και πώς θα αντιδράσουμε απέναντι στην κυβέρνηση της Κούβα. Έχω την αίσθηση εγώ ότι προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε τον διάλογο ανοιχτό, αλλά πρόκειται για μια χώρα η οποία δεν ακούει κανένα και συστηματικά παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριος Μακαμίλαν Σκότ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ισπανική Προεδρία και τις προηγούμενες Προεδρίες για τις προσπάθειες που κάνουν σε ένα πολύ σημαντικό τομέα. Χαίρομαι που εσείς, ε, Πρόεδρε, θα εμπλακείτε στις συζητήσεις οι οποίες θα ακολουθήσουν. Γνωρίζετε ότι μας ενδιαφέρουν όλα αυτά τα θέματα και ο Πρόεδρος Μπούζεκ μου ζήτησε σαν Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου να ασχοληθώ με τα θέματα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θέματα που παρακολουθώ εδώ και 20 χρόνια στα πλαίσια αυτής της Επιτροπής Υποεπιτροπής. Δύο σημεία. Το πρώτο, η θεσμική σχέση, η διοργανική μάλλον σχέση ανάμεσα ε, στο Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας και το ρόλο της ε, Άστον. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το Συμβούλιο να αναλάβει μια πιο αποφασιστική θα έλεγα θέση σε επίπεδο πολιτικό την οποία να στηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ ίδρυσα θα έλεγα την ε, Ευρωπαϊκή ε, Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, χρειάζεται να ξεφύγει λίγο από τα τετριμένα και να προχωρήσει σε θέματα μεγαλύτερο φιλόδοξα και σε σχέση με τη δημοκρατία, να μην φοβόμαστε τη λέξη της δημοκρατίας, ιδιαίτερα μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου τον μήνα Δεκέμβριο που ασχολήθηκε με το θέμα αν και δεν κατέληξε σε μια κάποια συνένεση. Η ατιμορρησία. Χαίρομαι που βλέπω στις προτεραιότητες της Προεδρίας τη λέξη αυτή. Νομίζω ότι θα πρέπει να φτιάξει ένα κατάλογο ατιμορρησίας εισαγωγικά το λέω αυτό για να ασχοληθούμε ε, με τα θύματα των, της τρομοκρατίας ε, και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκόσμια. Ξέρουμε ότι και στην Κίνα υπάρχουν παραβιάσεις ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ Πρόεδρε για την υπομονή σας. Αυτός ο κατάλογος για την ατιμορρησία θα έλεγα είναι πολύ σημαντικό. Ο Μάνφρεντ Νόβακ, υπεύθυνο για τα βασανιστήρια, μας είπε ότι αυτό το οποίο οι φυλακισμένοι ε, ικανοποιούνται αυτό από το οποίο είναι να κατονομαστεί ο αστυνομικός ή ο αξιωματούχος ο οποίος τους χτύπησε και ελπίζουμε κάποια στιγμή το Διεθνές Δικαστήριο να τους καταδικάζει. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπολσκι. Όχι, ο κύριος Όμπολς έχει το λόγο. Ε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Ισπανική Προεδρία. Μας παρουσίασε ένα πλήρες πρόγραμμα, ένα οδικό χάρτη, θα έλεγα πλήρη, γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν ε, και μεγάλη σε μέγεθος, θα έλεγα, η παρουσίαση των, του Ισπανού και νομίζω ότι αυτό πρέπει να μας ικανοποιεί. Έχουμε ένα συγκεκριμένο κατάλογο λοιπόν θεμάτων στα οποία μπορούμε να προχωρήσουμε. Η ανταλλαγή απόψεων την οποία θα κάνουμε από εδώ και πέρα θα είναι θετική στο βαθμό που θα μπορέσουμε βέβαια να συνεισφέρουμε και εμείς με επιμέρους ρυθμίσεις. Πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να έλθω σε τρία στοιχεία. Τρία στοιχεία τα οποία ίσως δεν ήταν, θα έλεγα, στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων που εξέθεσε ο αντιπρόσωπος της Προεδρίας. Έχουμε μία ολόκληρη σειρά από προβλήματα πάρα πολύ σοβαρά τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Προβλήματα τα οποία απαιτούν να υπάρχει μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Πρόκειται για προβλήματα, για περιπτώσεις που συνδέονται με φαινόμενα όπως η μετανάστευση, τα αιτήματα χορήγησης ασύλου, γενικά προσφύγων κτλ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ισπανική Προεδρία θα πρέπει να προσπαθήσει να διαχειριστεί εδώ ένα νέο κεφάλαιο του, ε, της συνθήκης της Λισαβόνα σχετικά με το δικαίωμα στη χορήγηση ασύλου. Και έχουμε να κάνουμε επίσης και με ένα κοινό σύστημα διαχείρισης εξωτερικών συνόρων. Όλα αυτά είναι καινοτομίε οι οποίες θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Το λέω αυτό γιατί πιστεύω προσωπικά ότι το θέμα έχει πολύ σημασία και θα πρέπει να τύχει μεγαλύτερης προσοχή. Σας διακόπτει ε, ε, κύριε Όμπολς λέει η πρόεδρος. Δεν έχουμε χρόνο, έχετε δύο λεπτά για να κλείσετε παρακαλώ. Είναι δύσκολο να κλείσω σε τόσο σύντομο χρόνο λέει ο κύριος Ομπιόλς. Κοιτάξτε, ακούσαμε μία παρουσίαση η οποία κράτησε πάρα πολύ ώρα, λέει ο κύριος Όμπιολς. Οι παρατηρήσεις λοιπόν σε δύο λεπτά σε μία τόσο μεγάλη ε, παρέμβαση ε, είναι περίπου αδύνατες. Γι' αυτό σας ζητώ να είστε υπομονετικοί μαζί μου, λέει αργά ο κύριος Ομπιόλς. Λοιπόν, συνεργασία και διάλογος με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών όπως επίσης και με όλες τις μη κρατικέ δομές είτε σε εθνικό, είτε σε κοινωνικό, είτε σε ε, διεθνές επίπεδο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η κοινωνία των πολιτών είναι πολύτιμο σύμμαχος και χρειαζόμαστε πιο συγκεκριμένους προσανατολισμούς για τη συνεργασία μαζί της. Επανέρχομαι στην βασική σας προτεραιότητα, κύριε Κουαδράδος, την καταπολέμηση της ε, θανατικής καταδίκης είναι σαφές ότι εδώ πρέπει να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις γιατί πράγματι έχουμε πάρα πολύ σωστά και καλά νέα από κάποιες περιπτώσεις, από κάποιες χώρες. Από την άλλη όμως, όπως είπε ο κ. Κουαδράδος, υπάρχουν και πάρα πολλοί δισταγμοί σε ορισμένες άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε συμμαχίες για να προχωρήσουμε στην ε, σωστή συνεργασία. Ε, κοιτάξτε, προσπαθήστε να κλείσετε, ξαναλέει η Πρόεδρος, τον κύριο Μπιόλς. Δε, δεν πειράζει, σταματώ λέει ο κ. Σομπιόλς. Λοιπόν, άλλοι οκτώ έχουν ζητήσει το λόγο. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σεβαστείτε τα δύο λεπτά που προβλέπονται για τον καθένα. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό σημείο να συζητήσουμε αμέσω μετά. Η κυρία Αντρεβική είναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Ισπανική Προεδρία για το γεγονό ότι μα ενημέρωσε σε σχέση με τι προτεραιότητε τη. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία ε, που έχει ε, το, το τι ακριβώς θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη σε διάφορα διεθνή φόρα για παράδειγμα στο Διεθνέ Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Υπήρχε πέρυσι, για παράδειγμα, μια ε, μεγάλη ε, διαφορά απόψε μεταξύ των κρατών μελών, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την έκθεση Κόρστοβα. Οπότε ε, ε συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπατε. Χθε, εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είχαμε μια ακρόαση για την Κούβα, δηλαδή την προώθηση τη δημοκρατία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί. εγώ αναφέρομαι ε, σε μια ε, πολύ πρόσφατη ανακοίνωση από τη Μαδρίτη ότι η Ισπανία υποστήριξε την ε, πρόταση ε, για σύναψη διμερού συμφωνία με την Κούβα και είπατε ότι ε, τώρα θα, μέσα στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών θα ασκήσετε πιέσει ε, στην Κούβα για να υιοθετήσει διατάξει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώ λοιπόν θα επιτύχετε μια ομοφωνία μεταξύ των κρατομελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώ θα πείσετε για παράδειγμα χώρε όπω η Τσεχία, οι οποίε είναι πολύ απρόθυμε να προβούν σε μια τέτοια συμφωνία με την Κούβα. Επίση, σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ εμπορικών συμφωνιών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεωρείται πω τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να αποτελούν ρήτρα σε όλα τα σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες γιατί υπάρχουν μια σειρά από συμφωνίες αυτού του είδους ε, προς κύρωση ε, και κατά την ακρόαση του κυρίου του ψήφου επιτρόπου κ. Ντεγκούχτε τέθηκε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε ήταν πολύ αποτελεσματικά, πολύ περιεκτικά αυτά τα δύο λεπτά της παρέμβασής σας. Θα ήθελα να πω πως αυτή η ακρόαση για την ε, Κούβα που έγινε κυρίως υπό την Αιγύρια του ΕΛΚ ε, συμμετείχαν οι δύο, άτομα από τα οποία έχουν λάβει το βραβείο Ζαχάροφ από την ίδια την Κούβα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, επόμενη ομιλήτρια κυρία Γκόμας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τον κύριο Κογιάδο για την ε, εξαιρετική παρουσίαση και σε σχέση με τις ε, προτεραιότητες που έχει θέσει στον εαυτό της η Ισπανική Προεδρία να πω ότι μπορώ μόνο να συμφωνήσω με αυτές. Νομίζω δηλαδή πως η, η σχέση την οποία αναφέρατε σε ό,τι αφορά την ισότητα των δύο φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το γεγονό ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των ε, ε, παιδιών σε ε, πόλεμε σειράξει ή το δικαίωμα σε πόσιμο νερό. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά και νομίζω πως ε, σε ό,τι αφορά την τήρηση τέτοιων, ε, το σεβασμό τέτοιων δικαιωμάτων, ε, κοινωνικών, πολιτισμικών και ούτω καθεξής, είμαστε πρωτοπόροι και δεν θα πρέπει να, είμαστε, να λαμβάνουμε μια αμυντική στάση όταν πολεμάμε για τέτοια ανθρώπινα δικαιώματα. Και συμφωνώ με αυτό που είπε η Αμνηστία, ότι δηλαδή η στάση που θα τηρήσουμε απέναντι στην έκθεση Κόρσταν θα είναι καθοριστική για το τι θα κάνουμε εμείς. Δηλαδή, στο πλαίσιο και της συνδίκης της Λισαβόνας θα είναι σημαντική σημαντικό να υπάρχει μια καλή σχέση μεταξύ των όσων εκπροσωπεί ε, προς τα έξω Ευρωπαϊκή Ένωση ως προ τα ανθρώπινα δικαιώματα και ως προς το τι πράττει σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της. Είναι λοιπόν θεμελιώδου σημασία και στο πλαίσιο της, ε, του αγώνα για την καταπολέμηση των βασανιστήριων ε, και στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας να το τηρήσουμε αυτό ή για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ανάληψη των εθνών. τα, εκείνα τα renditions, εκείνες οι εκδόσεις δηλαδή που γινόταν από την ε, κυβέρνηση Bush. Ε, και είχαμε για παράδειγμα εκεί ε, Πολωνία και Ρουμανία ως χώρες οι οποίες είχαν συνεργαστεί αλλά όχι μόνο νέα κράτη-μέλη και παλαιά κράτη-μέλη. Η Γερμανία για παράδειγμα είναι σίγουρο πως είχε συνεργαστεί. Μετά, σε ό,τι αφορά την πολιτική γειτονία. Και εκεί είναι πολύ σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για παράδειγμα, σε σχέση με το Μαρόκο. Στο πλαίσιο τη αναπτυξιακή πολιτική και στο πλαίσιο και των σχέσεων με την Αφρικανική Ένωση, είναι και πάλι σημαντικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί και εκεί πάντα προσπαθούμε να δώσουμε έμφαση. Αυτά να τα να τους δώσουμε προτεραιότητα και να παραβέμψουμε εδώ και στην περίπτωση του Σουδάν και στο ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή εκεί. Ε, για παράδειγμα, μια γυναίκα η οποία ήταν αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, συνελήφθη στην Αιθιοπία και εμείς ε, παρέχουμε υποστήριξη σε αυτή τη χώρα. Να καλωσορίσω τον Ισπανό συνάδελφο. Αυτά τα οποία είπε ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε τις προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές και να μην αζητήσουμε την εφεύρεση νέων, αυτό είναι κάτι που με βρίσκει σύμφωνα όπως επίσης και αυτά τα οποία είπατε για την διάσκεψη για τους ομοφιλόφιλους και τους φιλομεταβατικούς και αυτό είναι ένα καλό νέο και θα ήθελα να συμφωνήσω και με αυτά τα οποία έχει πει η Amnesty International για ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα να δω επίσης τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε επίπεδο των νέων δομών για την εξωτερική πολιτική η κάθε άστον θα μας διαβουλεύετε σαν κοινοβούλιο, αλλά θα έχετε και εσείς συζητήσεις ε, μέσα στο Συμβούλιο, θα πρέπει ε, να ε, μας ενημερώνετε σωστά. Έχει σημασία το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, διότι μέχρι τώρα τα πράγματα πήγαν σχετικά καλά, αλλά σε κάποια περιορισμένη εμβέλεια θα έλεγα η παρέμβασή μας ήταν αποτελεσματική δηλαδή σε συγκεκριμένους λίγους τομείς. Δεύτερον, ξέρω ότι δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για τον κώδικα συμπεριφοράς, για τους αναπήρους. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Το θέμα είναι να ελέγξουμε τις νέες πολιτικές και τα νέα προγράμματα έτσι ώστε να γίνονται σεβαστά το περιεχόμενο και οι ρήτρες ε, της σύμβασης αυτές. και οι απειλές, η αντιμετώπιση των απειλών για την θανάτωση των ομοφιλοφίλων ανδρών και γυναικών στην Ουγκάντα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε από πολύ κοντά. Η Amnesty International για όλα αυτά έχει κάνει συγκεκριμένες δηλώσεις. Το θέμα είναι να δούμε ε, τι γίνεται και στη Λωρίδα της Γάζα και δεν είναι θέμα ε, γενικότερα εξωτερικής πολιτικής ή ευρωπαϊκής ενότητας αλλά είναι θέμα σεβασμού των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζα και δεν θα πρέπει εδώ να βρίσκουμε ε, άλοθη στο ότι δεν είμαστε ενωμένοι γύρω από την αντιμετώπιση του Μεσανατολικού. Ευχαριστώ πολύ. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο σας είχα πει προηγουμένως. Ξέρετε ότι στον τύπο λέγεται ότι η Ουγγάντα από ό,τι φαίνεται απέσυρε την πρόταση νόμου η οποία καταδίκαζε σε θάνατο υποτίθεται τους ομοφιλόφιλους. Αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο. Λοιπόν, επόμενη ομιλήτρια. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη σχετικά με την προάσπιση αυτών που προασπίζονται με τη σειρά του τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ξέρουμε τι γίνεται στο Ιράν, ε, μέλη της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφοι. Δεν είναι δηλαδή απλά ε, άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά δεν πάβουν να καταγγέλουν με ελεύθερες φωνές το τι κάνει η κυβέρνηση εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτούς, να τους βοηθήσουμε δηλαδή. Και η άλλη ερώτησή μου αφορά την ε, επιρροή του διαδικτύου στα ανθρώπινα δικαιώματα. Βλέπετε κάποιες δυνατότητες εκεί. Ευχαριστώ κυρία Σάκε. Danke, frau Vorsitzende. ich werde nicht ausschweifend reden aber es ist eigentlich unmöglich Είναι αδύνατο να συζητήσει κανείς μια έκθεση 89 σελίδων. Δική μας δουλειά είναι να κάνουμε προτάσεις και να δίνουμε ιδέες. Πρώτη παρατήρηση για την θανατική ποινή. Η Ισπανική Προεδρία είναι ιδιαίτερα στρατευμένη στο θέμα. Θα έπρεπε εμείς ως Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να ζητήσουμε και ένα ψήφισμα πω τον ΟΗΕ για την υποστήριξη του Γενικού Γραμματέα στον αγώνα για την κατάργηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάμε για δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν μιλάμε όμως για γεωγραφικές περιοχές και περιφέρειες δεν λέμε τίποτα. Λέμε ναι, εντάξει είναι πολύ σημαντικό αλλά αναπερίπτωση δεν λέμε τίποτα. Θα έπρεπε κάπως να ε, έχουμε άλλου είδους αναφορές σχετικά. Βία κατά των γυναικών Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι η Ισπανική Προεδρία αναλαμβάνει. Και γνωρίζω ότι έχει δημιουργηθεί ένα σημείο, ε, έχει υπάρχει μια πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί ένα σημείο επαφής ε, για ε, γυναίκες από τη Λατινική Αμερική, οι οποίες θα μπορούν να, να έρχονται σε επαφή, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιες αντιθέσει, οπότε θα ήθελα να γνωρίζω ποιε ακριβώ είναι οι αρχέ οι οποίε αντίθενται σε αυτό. Ε, εκείνο που αναφέρθηκε τώρα από συναδέλφους ε, σε σχέση με την λάθρο μετανάστευση ε, θα πρέπει η Frontex και άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες για τη φύλαξη των συνόρων να εργάζονται πάντα με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα ήθελα να ξέρω πώς θα το διασφαλίσει αυτό η Ισπανική Προεδρία. Επίσης, σε σχέση με τα βασανιστήρια Πού έχουμε φτάσει σε σχέση με τη συνεργασία των κυβερνήσεων για αυτά τα, τις μυστικές εκδόσεις των ε, υπόπτων, τα ε, renditions και ε, σε ό,τι αφορά και τη συνεργασία με το Διεθνές Επινικό Δικαστήριο. Και κυρία Πρόεδρε, τι ακριβώ μου προτείνετε τώρα, δηλαδή να συζητήσω απευθείας τι με την Ισπανική Προεδρία, δηλαδή ε, δεν ήξερα ότι στην Επιτροπή μας ε, έχουμε δικαίωμα μόνο να παίρνουμε το λόγο για δύο λεπτά ή τουλάχιστον να μας το λέτε αυτό από την αρχή. Ούτε κι εγώ ήξερα ότι η Ισπανική Προεδρία θα είχε να μας παρουσιάσει ένα τόσο λεπτόμερες πρόγραμμα και ότι θα χρειαστεί μισή ώρα για να το παρουσιάσει. Εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσουμε με τη συζήτησή μας. Και ε, πραγματικά θα ήθελα σας παρακαλέσω να συνεχίσετε να τηρείτε αυτά τα δύο λεπτά όλοι οι μελητές. Εν πάση περιπτώσει έτσι καλώ θα πάρουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Ο πρόεδρος τώρα έχει το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι η παρουσίαση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και μας ε, έδειξε ε, λεπτομερώς τις κατευθύνσεις που ακολουθεί η Ισπανική Προεδρία. Αλλά έχω να θέσω δύο ερωτήματα. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως ε, ε, τα καθήκοντα, για παράδειγμα αυτά που έχετε θέσει στον εαυτό δεν είναι καθήκοντα που αφορούν μόνο μια εξάμενη προεδρία, είναι μακροπρόθεσμη στόχη. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο ε, η Ισπανική κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας και η δική σας υπηρεσία η αρμόδια Εάν λοιπόν έχετε ε, επαφέ με τι αντίστοιχε υπηρεσίε ε, του Βελγίου και τη Ουγγαρία, αφού πρόκειται για τι επόμενε χώρε οι οποίε θα αναλάβουν την ε, Προεδρία του Συμβουλίου και κατά συνέπεια θα κληθούν να εφαρμόσουν αυτά τα, αυτούς τους στόχους. και το δεύτερο ερώτημα είναι πως τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν παρεμβάσεις σε συγκεκριμένε ε, περιπτώσει, όχι γενικού στόχου. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη σύλληψη στη Μόσχα τη κυρία Αλεξέγεβα, τι ακριβώ σκοπεύετε να κάνετε. Ή το ζήτημα του, Ευρωπαϊκού, του Ευρωβουλευτή ε, και το γεγονό ότι δεν του επιτράπει η είσοδο ε, στην Κούβα. Θα κάνετε κάτι συγκεκριμένο για αυτέ τι περιπτώσει. Köszönöm, romániai magyarként külön örvendek, hogy Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο σαν Ούγγρος από την Ρουμανία από το ότι οι επόμενες προεδρίες, η Ισπανική δηλαδή και οι επερχόμενες, η Βελγική και η Ουγγρική θα προσπαθήσουν συνεργαζόμενες από κοινού να αντιμετωπίσουν αυτή την δύσκολη μεταβατική περίοδο μία περίοδο η οποία ξεκίνησε μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Ισπανική Προεδρία διότι έχει βάλει στις βασικές της προτεραιότητες τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρόκειται για ευρωπαϊκές αλλά και όχι μόνο και διεθνείς καθολικές θα έλεγα μορφές ε, προτεραιότητας. Ξέρετε ότι ήδη στο τέλος του προηγούμενου χρόνου ε, καταλήξαμε σε μία απόφαση η οποία καταδικάζει γενικά ε, της θανατική ποινή, ιδιαίτερα μετά από τα επεισόδια στο Σινκιάνγκ και τις ε, παράδεκτες αντιδράσεις της κινέζικης κυβέρνησης. Ξέρουμε ότι οι περισσότερες εκτελέσεις γίνονται στην Κίνα και αφορούν κυρίως τους Ουιγούρους. Από την άλλη η κατάσταση σε άλλες χώρες έχει σχετικά βελτιωθεί. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το μορατόριο για τη θανατική ποινή στην Ρωσία και τουλάχιστον εκεί έχουμε θετικό σημείο. Πάντως το θέμα των μειονοτήτων γενικότερα δεν το άκουσα ιδιαίτερα από πλευρά της Ισπανικής Προεδρίας. Ξέρετε ότι οι εθνοτικές μειονότητες ε, είναι οι μεγαλύτεροι θα έλεγα κατηγορίες. Είναι, υπάρχουν εθνοτικές μειονότητες, γλωσσικές μειονότητες, θρησκευτικέ μειονότητες που υφίστανται διακρίσεις σε πάρα πολλές ε, περιοχές του κόσμου. Ζητώ λοιπόν να μου πει η Ισπανική Προεδρία τι μπορεί να κάνει έτσι ώστε και εδώ και στις τρίτες χώρες και αναφέρομαι κυρίως στις τέως κομμουνιστικές χώρες αλλά και τις σημερινές χώρες που παραμένουν κομμουνιστικές πώς θα γίνουν σεβαστές οι μειονότητες και πώς ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μειονοτήτων θα είναι προϋπόθεση για την πιθανή είσοδο κάποτε των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρομαι στη Σερβία και την Ουκρανία. Ευχαριστώ κύριε Τούκες. Τελευταίος συνάδελφος, Πρέρα. Και μετά θα ακούσουμε τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ για αυτά τα οποία είπατε για τη θανατική ποινή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ο εκπρόσωπος της, της Προεδρίας του Συμβουλίου είπε ότι θα δοθεί και συγκεκριμένη προσοχή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και γι' αυτό παρακαλώ να αναφερθώ σε μία την οποία ανέφερε και η κυρία Χάουταλα. Πρόκειται για μία περίπτωση η οποία θα έλεγα είναι παραδειγματική είναι η περίπτωση του Ξιαομπό. Ο ο Λίου Ξιαομπό, έχει καταδικαστεί σε 11 χρόνια στη φυλακή στην Κίνα στο τέλος Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ γιατί επανήλθατε σε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση, λέει η Πρόεδρος, και δίνω το λόγο τώρα στην Βερονή Καρνό από τη Γενική Διεύθυνση Ρελέξ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαίρομαι που είστε μαζί σας σήμερα και δεν ξέρω αν μπορείτε να σχολιάσετε την συζήτηση η οποία προηγήθηκε και την παρουσίαση της Ισπανικής Προεδρίας όπως και τη μεταβατική περίοδο την οποία διασχίζουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες οριζόντιες παρατηρήσεις για να συμπληρώσω αυτά τα οποία είπε ο Χουάν σχετικά με τη συνθήκη, τη Λισαβόνα. Πράγματι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Ο συνάδελφος της Άμνεστη είπε ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε τη θέση σας απέναντι σε όλους τους εταίρους σας. Θα πάρει χρόνο αυτό. Έχουμε δύο θα έλεγα στόχους. Πρώτον, να δείξουμε ότι έχουν υπάρξει αλλαγές στις εξωτερικές σχέσεις δεν υπάρχει Προεδρία, υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Και όπω είπε η Ισπανική Προεδρία, ομιλούμε πλέον εξ ονόματο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του υπάτου εκπροσώπου. Ε, κάτι το συμβολικό, ίσως το παρατηρήσατε, ιδιαίτερα που είναι πολύ θετικό για παλιούς υπαλλήλου όπως εγώ. Την 16η Ιανουαρίου για πρώτη φορά στην συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπήρχε ένα ταμπελάκι στην τράπεζα που έλεγε Ευρωπαϊκή Ένωση και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε και τη δήλωση για το Αφγανιστάν. Συμβολικό σε αυτή τη φάση αλλά αρκετά σημαντικό. Έχουμε λοιπόν την υποχρέωση να δείξουμε προς τα έξω κάποιες αλλαγές. Έχουμε όμως και μια υποχρέωση να διασφαλίσουμε την συνέχεια των ρυθμίσεων. Είναι αλήθεια ότι θα πηγαίνουμε ψάχνοντας ώσπου να έχουμε στη διάθεσή μας ε, μια πλήρως λειτουργούσα εξωτερική υπηρεσία. Έχουμε πραγματιστικούς στόχους σε συνεργασία με την Ισπανική Προεδρία, τα πράγματα πηγαίνουν καλά και έχει σημασία να δείξουμε ότι χρησιμοποιούμε όλοι ε, τον ίδιο λόγο. Είναι σαφές ότι θα απλοποιηθούν τα πράγματα και σε σχέση με τις τρίτες χώρες δεν θα υπάρχουν τρόικα πλέον, αλλά από την άλλη είναι αλήθεια ότι η Ισπανία που έχει συγκεκριμένες ευθύνε θα υποστηριχθεί από τη Γενική Γραμματεία και της Ευρωπαϊκής, του Συμβουλίου συγγνώμη, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά έχουν μια κάποια σημασία. Λόγω του ότι λοιπόν διευκρινίζονται προοδευτικά οι δομές και αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μας την τελική μορφή της εξωτερικής υπηρεσίας, τότε θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με πλήρως, ε, θα έλεγα, αποτελεσματικό τρόπο. Οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διάφορες χώρες είναι, θα έλεγα, εγκατεστημένες ε, με καλό τρόπο. Υπάρχουν περίπου 50 ε, αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκπροσωπούν τώρα πλήρως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις υπόλοιπες βρισκόμαστε σε μεταβατική φάση. Όπως είπε ο συνάδελφος, η κατάσταση των αντιπροσωπιών αυτών και η θέση τους στους διεθνείς οργανισμούς είναι κάτι το πιο ευαίσθητο και εκεί η διαδικασία μετάφασης θα πάρει περισσότερο χρόνο. Ήδη στη Νέα Υόρκη υπάρχει ένα σαφές σύστημα ρυθμίσεων, ρεαλιστικών λύσεων, που συνδέει θα έλεγα αυτούς οι οποίοι υπάρχουν στη Νέα Υόρκη και συνδέει επίσης τις υπηρεσίες γενικότερα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και την υπηρεσία της υπάτης εκπροσώπου. Ήδη έχουν γίνει κάποιες προκαταρτικές συναντήσεις και υπάρχει μια μεγάλη ευαισθησία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι προσπάθειές σας όπως και οι προσπάθειες των συναδέλφων σας για να απογκαιτοποιήσουμε σε εισαγωγικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και για να αντακαταστήσουμε μια βασική ανησυχία και αυτά τα οποία προσπαθούμε να τα κάνουμε έτσι και αλλιώς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι το οποίο θα μας ικανοποιήσει. Όπως είπε η κυρία Άστον, σε δύο είναι οι βασικές αρχές. Πραγματισμός από τη μία, αποτελεσματικότητα από την άλλη. Ένα μέγεθος για όλους δεν ισχύει πια, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την δημόσια διπλωματία. Μια άλλη παρατήρηση που καλύπτει κάποιες ερωτήσεις αφορά την κοινωνία των πολιτών. Έχω την εντύπωση ότι η κοινωνία των πολιτών πρέπει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Γνωρίζετε ότι σε σχέση με τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα συστηματικά προσπαθούμε να οργανώνουμε είτε ειδικά σεμινάρια είτε κάποιες μορφές διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών που οργανώνονται από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ξέρω ότι ορισμένα μέλη της υποεπιτροπής σας, Πρόεδρε, θα ασχοληθείτε στην ε, συνάντηση που προβλέπετε να γίνει με την κοινωνία των πολιτών στη Ρωσία. Αυτό είναι απαραίτητο, μιας και μιλάμε αρκετά για τη Ρωσία. Υπάρχει κάτι το θετικό, όχι για πρώτη φορά, έχουν προηγηθεί και άλλες θετικές. Με το νέο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης θεωρούμε ότι η Ρωσία θα υιοθετήσει το 14ο πρωτόκολλο του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα συνδεθεί πλέον με την Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Δεν μιλάω για νομική ρύθμιση απλά, αλλά καλό θα είναι στην γειτονία μας, στην πολιτική, να υπάρξουν κάποια θετικά βήματα. Πάντα γύρω από την κοινωνία των πολιτών και σε σχέση με τον Κάφκασο και τη Βόρειο Αφρική και την ε, Αφρικανική Ένωση έχουμε συγκεκριμένες μορφές διαλόγου οι οποίες εξελίσσονται και καλύπτουν κάποιες από τις ανάγκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντίθετα με αυτά τα οποία ακούστηκαν υπάρχουν ξεκάθαρες οδηγίες για τις διπλωματικές μας αντιπροσωπείες είτε της τέος της Επιτροπής είτε των κρατών μελών για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτούς οι οποίοι προασπίζονται ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε αυτά τα σημεία επαφής, τα focal points. Τα πράγματα δηλαδή εξελίσσονται. Ένα άλλο πράγμα σχετικά με την συνοχή που πρέπει να μας χαρακτηρίζει εσωτερικά και εξωτερικά. Το είπαν και πολλοί συνάδελφοί σας. Είναι μια πρόκληση ολοένα και πιο μεγάλη αυτή. Αναφέρθηκαν πάρα πολλά στοιχεία. Ακούσαμε ότι για τα βασανιστήρια και για κάποια άλλα σχετικά θέματα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κάνουν ιδιαίτερες προσπάθειες. Είπαμε επίσης ότι και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν συγκεκριμένες προσπάθειες. Για τις γυναίκες αναφερθήκαμε στη μεγάλη σημασία που έχει το 2010 και ελπίζουμε ότι η κυρία Ρέντινγκ που είναι πλέον ε, σε εσωτερικό επίπεδο η Επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα να πάρει μέρος στη συνάντηση τον Μάρτιο για την κατάσταση των γυναικών. Όλα αυτά τα λέω για να διευκρινίσω ότι από πλευρά των θεσμικών οργάνων γίνεται μια προσπάθεια για μεγαλύτερη συνοχή, γιατί αμφισβητείται όλο και περισσότερο η αξιοπιστία μας. Υπάρχουν και τα θέματα της μετανάστευσης και εκεί υπάρχουν δύο ανοιχτά προβλήματα. Το πρώτο θα το αντιμετωπίσετε στα πλαίσια του hearing για αυτούς που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί η πολιτική μας είναι δραστήρια και υπάρχει και το θέμα των θεωρήσεων. Εκεί τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα και κάθε φορά πρέπει να καταλήγουμε σε συγκεκριμένες λύσεις. Σχετικά με τη διαφάνεια και την ανοιχτή διπλωματία, με τη Σουηδική Προεδρία όλοι επικυρώσαμε τις νέες κατευθυντήριες πολιτικές γραμμές και νομίζω ότι η Ισπανική Προεδρία θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση. Οργανώνουμε το Μάρτιο κάτι γύρω από αυτό για να συνεχίσουμε να δείχνουμε ότι σε επίπεδο διαφάνειας αυτού το οποίο κάνουμε δεν θα σταματήσουμε. Η ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οποία δημοσιεύουμε μαζί με το Συμβούλιο, θα τεθεί προσυζήτηση σύντομα και θα συμβάλλει στην πολιτική της διαφάνειας. Ο κ. Μακμίλαν Σκοτ λυπήθηκε γιατί ε, η λέξη δημοκρατία δεν είναι ανάμεσα στις προτεραιότητές μας. Δεν μπορούμε να βάλουμε τα πάντα. Προφανώς δεν υπάρχει απλά μια συμβατική συμφωνία θα έλεγα για τη δημοκρατία, αλλά το Συμβούλιο μας έχει δώσει μια ξεκάθαρη εντολή έτσι ώστε να ορίσουμε κάποιες πιλωτικές χώρες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να ολοκληρώσουμε την πολιτική μας για τη δημοκρατία. Νομίζω λοιπόν ότι η Ισπανική Προεδρία ή εν πάση περιπτώσει εξ ονόματος ε, της, ε, είπα, εκπροσώπου θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Σπίλμπαγκ και όλους τους συναδέλφους που ε, Πίμπαλξ και με όλους τους συναδέλφους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Τώρα, γιατί υπάρχουν κάποιες ε, αντιφάσεις και γιατί δεν μπορούμε να συνδυάσουμε όλα τα συμφέροντα. Η απάντηση είναι ότι πράγματι υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις σε επίπεδο ε, συνοχής, αλλά δεν μπορούμε να τα αναμίξουμε όλα σε επίπεδο τυπικό αν θέλετε επίσημο έχει διασφαλιστεί μια κάποια μορφή συσχετισμού των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου, των εμπορικών συμφωνιών που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση μάλιστα οι περισσότερες και των συμφωνιών συνεργασίας, εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτές είναι συμφωνίες που ε, γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευση σε διαφορετική βάση στις εταιρικές συμφωνίες. Υπάρχουν πάρα πολλές ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Με τις χώρες της Ασίας έχουμε αρκετές δυσκολίες για τη διαπραγμάτευση αυτών των συμφωνιών, αλλά εμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και υπάρχει μια γέφυρα θα έλεγα ανάμεσα στις ε, πολιτικές συμφωνίες και στις εμπορικές συμφωνίες. Αυτό το οποίο θα πρέπει κυρίως να γίνει είναι να διαβουλευτούμε μεταξύ μας εκ των προτέρων και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις μορφές συνοχής. Με το GSP Plus προχωρήσαμε προς τον στόχο της διαφάνειας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα αυτό ε, για να το θεωρήσουμε σαν ένα κίνητρο και για τις εμπορικές συμφωνίες έτσι ώστε οι χώρες με τις οποίες συνάπτουμε τις συμφωνίες να σέβονται καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ε, συνδικαλιστικές ελευθερίες. Για την πολιτική γειτονία κάνουμε αρκετά πράγματα. Το μέσο για την γειτονία και οι αιτήσει εκθέσει υπογραμμίζουν συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό δεν μα κάνει μόνο φίλου. Το Μαρόκο αναφέρθηκε επίσης. Το Μαρόκο είναι μια χώρα η οποία είναι συνδεδεμένη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε πολλές ελπίδες για να είναι πρότυπο για τις χώρες της Μεσογείου και τις αραβικές χώρες σχετικά με την κριτική που ασχεί η ο, ο Μακμίλαν Σκότ. Νομίζω ότι οι συζητήσεις που θα γίνουν στο μέλλον δείχνουν ότι τα πράγματα έχουν ξεκινήσει και εξελίσσονται πια. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες αρκετά γραφειοκρατικές και λυπάμαι γι' αυτό και ελπίζω το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν αναθεωρήσουν τον οικονομικό κανονισμό, να μας δώσουν κάποια μέσα έτσι ώστε να δράσουμε ταχύτερα. Ελπίζω, λέει η κυρία Χούταλα, η συνεργασία μας να συνεχιστεί. Η συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή και σε εσάς, στη δική μας Επιτροπή και σε εσά ήταν πάντα θετική. Θα περάσουμε τώρα στον εκπρόσωπο της Ισπανικής Προεδρίας και βέβαια έχουμε κάποια προβλήματα με το ωράριο εργασίας μας. Θα ήθελα όμως να δώσω το λόγο στον, στον εκπρόσωπο της Προεδρίας να αντιδράσει στις παρατηρήσεις των συναδέλφων μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας η Ισπανία έχει μακρόχρονη και θλιβερή εμπειρία με θέματα τρομοκρατίας. και σας ευχαριστώ για την πρότασή σας. Θα ληφθεί υπόψη στις, στον εξωτερικό μας διάλογο. Τώρα για την Κούβα. Ψύχρολουσία οι διαπραγματεύσεις μας με την Κούβα. και σίγουρα όπως ε, είπε και ο Υπουργός Εξωτερικών θα θέλουμε να ξεπεράσουμε το επίπεδο των διαβουλεύσεων που έχουμε μέχρι σήμερα αλλά γι' αυτό χρειάζεται η συνένεση των 27 και για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα δούμε αν η πολιτική κατάσταση θα μας το επιτρέψει και κάποιος άλλος ανέφερε την Κούβα υπάρχει συγκεκριμένη διαχείριση για την ελευθερία της έκφρασης ε, και της τεχνολογίας διότι το σύστημα των blog είναι πολύ σημαντικό για την έκφραση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα Τώρα για τον κύριο Μακμίλαν, η Βερονή Καρνό το είπε. Εμείς είπαμε να ξαναδραστηριοποιήσουμε ε, την Task Force για την Δημοκρατία. Κύριε Μπιόλς, είμαι στη διάθεσή σας για το θέμα της μετανάστευσης είναι θεμελιώδες. Χρειάζεται συνέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απ' έξω και από μέσα. Ε, αυτό το λέμε συνεχώς στις διαπραγματεύσεις μας. Αλλά πριν ε, διαπραγματευτούμε πρέπει να έχουμε λύσει και τα προβλήματα μέσα στην Ένωση. Είχαμε επίσης και διαβουλεύσεις, ένα γύρο διαβουλεύσεων εδώ στις Βρυξέλλες και στη Μαδρίτη με την κοινωνία των πολιτών. Εμείς θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των προσώπων. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ατιμορρησία. Εμπορικές συμφωνίες. Παράδειγμα, η Σρι Λάνκα. Εμείς ε, θα έχουμε μία προσωρινή <coughs> ανάκληση των σχέσεών μας με τη Σρι Για το Μαρόκο έχουμε αυτό το θλιβερό παράδειγμα της Χαϊδάρ. Τώρα για... θα ήθελα να μου αναφέρετε για το Σουδάν τη συγκεκριμένη περίπτωση και για την Αιθιοπία που βρίσκεται επίσης στο κείμενο της αμνηστίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή τη χώρα θα ενέκρινε μια ενιαία εντολή. Κύριε Χάουιτ, σας ευχαριστώ. για τα προβλήματα της φιλομεταβατικότητας και του LGBT. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Το ετήσιο σχέδιο θα παρουσιαστεί το Μάιο στο πιο ψηλό επίπεδο, δηλαδή ελπίζουμε να έρθει ο Υπουργός να το παρουσιάσει. Είπαμε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι επιμελή και στο εσωτερικό τους. Και το μέσο επικύρωσης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Για το Ιράκ, ε, οι ε, δημοσιογράφοι και αγωνιστές, ε, στο Ιράν, συγγνώμη, αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δημοσιογράφοι, ναι, θα στείλουμε συγκεκριμένες προτάσεις και στο Ιράν για να μπορέσουμε να έχουμε και διαπραγματεύσεις εδώ στις Βρυξέλλες. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Πρέπει να το δούμε μέσα από μια πολιτική προοπτική. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση προεμφυλίου πολέμου. και θα κοιτάξουμε να μην περάσει η υποψηφιότητα του Ιράν για το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κύριε Βιλάν, για την θανατική ποινή. Εμείς ντρεπόμαστε πολλές φορές όταν πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε τρίτες χώρες ε, για πράγματα τα οποία εμείς δεν έχουμε υλοποιήσει μέσα στην Ένωση. Τώρα στο κόμμα ε, έγινε μια ευγενική υπόμνηση σε κράτη-μέλη για τα πράγματα που έχουν παραμελήσει στις χώρες τους. Μία από τις στρατηγικές της Προεδρίας για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τους αγωνιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι να προσπαθήσουμε μέσα από αιτήσεις συνεδριάσεις να δούμε πού λείπει αυτό το κομιτέ τελειεζόν για να το φτιάξουμε. Χρειάζεται όμως πάντα να έχουμε έναν σύνδεσμο ανεξαρτήτως εθνικότητας, έναν σύνδεσμο στις τρίτες χώρες. Κύριε Σέμκι, Έχουμε στενή συνεργασία με το Βέλγιο εδώ και, πολλούς μήνες, μερικούς μήνες. για το τι θα πρέπει να προετοιμάσουμε ε, τους επόμενους ε, μήνες ε, και έχουμε και μία Ουγγαρέζα υπάλληλο η οποία εργάζεται στο Υπουργείο στην Ισπανία για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να μπορέσουμε να συντονιστούμε σε αυτές τις περιπτώσεις κυρίως δε στα θέματα πράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε χώρες όπως η Ρωσία και θέλουμε μορατόριουμ ε, της θανατικής ποινής και θα έχουμε και μία δήλωση για το μορατόριουμ της θανατικής ποινής στην Εβάδα. Η πρώτη δήλωση που έγινε από την εκπρόσωπο αυτή τη βδομάδα ήταν η δήλωση για την κοινότητα Μπαχάη στο Ιράν. Υπάρχουν ελάχιστα σημεία τα οποία δεν θίξατε. Νομίζω ότι απαντήσατε τάχιστα σε όλα όσα έγιναν. Ε, είχαμε και όμως και μία ερώτηση για την ανταλλαγή εχμαλώτων. Ήταν σαφής η ερώτηση. και οι απαγωγές ε, επίσης ε, των κρατουμένων. Ε, Εκτιμώ το όσα είπατε. Αλλά δεν αναφερθήκατε και στο ζήτημα της εξωτερικής μας υπηρεσίας, δηλαδή της αρμόδιας για τις συνεργασία στις εξωτερικές υποθέσεις. Πρόεδρο. Ε, κύριε Χάουαρντ, θα ήθελα να επανέλθουμε σε αυτά τα ζητήματα με την Ισπανική Προεδρία και ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον Ευρωπαϊκό ε, στο πλαίσιο τη εξωτερική πολιτική, γιατί πραγματικά δεν έχουμε χρόνο. Αλλά αν θέλει ο κύριο Σεντουάρντι να πει κάτι σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Κύριο Χάουαρντ, θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε έστω και μια δήλωση δέσμευση από πλευρά τη Ισπανική Προεδρία για ένα μόνο λεπτό. Γιατί αυτό αποφασίστηκε από την ομάδα μα και έχουμε και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εδώ. Δηλαδή δεν θέλετε να περιμένετε, λέει η πρόεδρο, στις 25 Ιανουαρίου, γιατί εμεί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Σα λέω ότι έχουμε καθυστερήσει 45 λεπτά και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν για να ξεκινήσει η ακρόαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία. Σας ζητώ συγγνώμη δηλαδή, αλλά πραγματικά έχουμε φτάσει σε ένα Ωραίο εδώ. Έχουμε, πολύ περιορισμένο χρόνο. απευθύνω μια έκκληση να επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα το συντομότερο δυνατό. Ε, να... Δεν μπόρεσα να απαντήσω σε όλα. Τώρα θα πρέπει να συντονιστούμε με τα αρμόδια όργανα για τις απαγωγές, ε, για τις πτήσεις της CIA. το ψάχνουμε σε εθνικό επίπεδο για το ποιο θα είναι αυτός που θα πρέπει να απολογηθεί. Και θα το συζητήσουμε στις 29 Ιανουαρίου με τις, ε, στις διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Τώρα για τις ανταλλαγές δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα. Βέβαια το Βέλγιο δεν είναι απαραίτητα παρόν σε αυτόν τον διάλογο αλλά θέλουμε να το ξεκαθαρίσουμε αν θα έρθει ή όχι. Εμείς θεωρήσαμε ότι στην ημερήσια διάταξη της κόμμα θα δίνουμε και όλα τα στοιχεία, τα ενημερωτικά στοιχεία που χρειάζονται στα κράτη-μέλη. Και υπάρχουν και διαφορετικοί όροι μεταξύ Νέας Υόρκης και Γενέβης. Έχουμε, στη Νέα Υόρκη έχουμε ένα joint team το οποίο εργάζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενώ στη Γενέβη δεν καταφέραμε να έχουμε αυτό το joint team ε, Νομίζω ότι η Νέα Υόρκη μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσουμε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο και να εφαρμόσουμε δηλαδή και τη Λισαβόνα. Ευχαριστώ την Ισπανική Προεδρία για αυτή την παρουσίαση και για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που μίλησαν. Λοιπόν, Βρισκόμαστε στην αρχή της Ισπανικής Προεδρίας και θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε σε διάφορα θέματα της Ισπανικής Προεδρίας κατά τους επόμενους έξι μήνες. Προτείνω να πάμε στο σημείο 4 που αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα στην Συρία, κυρίως στο πλαίσιο της επικείμενης συμφωνίας μεταξύ Συρίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Μινίκ Μποντί είναι ο σχετικός εισηγητής αλλά η πτήση του έχει καθυστέρηση και δεν θα μπορέσουμε να τον ακούσουμε. Κυρία Πρόεδρε, εγώ εδώ είμαι. Ο Μάριο Νταβίτ χρειάστηκε να φύγει. Α, ο Μάριο Νταβίτ χρειάστηκε να φύγει, μάλιστα. Euh, που είναι πρόεδρος της αντιπροσωπείας ε, του Μασρέκ. Συγγνώμη κύριε Μποντίσια ε, για το λάθος. Γι' αυτό το σημείο θα μιλήσουν διάφοροι, ο Μάρκ Σάντεν Πούτσεν, το Ευρωμεσογειακό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η κυρία Νασίρα Ιου Μπουλεβάτ για την Κομισιόν και είναι παρούσα σε περίπτωση ερωτήσεων. Καλέσαμε και την Συριανή αντιπρεσβεία ε, η οποία δεν ήρθε και φυσικά δεν μας απάντησε. Δεν μας είπε ούτε θα έρθω ούτε δεν θα έρθω. Συγγνώμη για το λάθος και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που με καλέσατε στην Επιτροπή σας για να σας αναφέρω το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία και πιο συγκεκριμένα υπό την προπτική σύνδεσης. Πόσο χρόνο μου δίνετε κυρία Πρόεδρε? Πόσο χρόνο μου δίνετε κυρία Πρόεδρε? Πέντε λεπτά έχετε κύριε Μποντής. Δεν θα τα καταχραστώ, λέει ο κύριος Μποντής. Η κατάσταση των ανθρωπίνων στη Συρία θα πρέπει να εξεταστεί από τέσσερις πλευρές. Πρώτο, το θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιφερειακό πλαίσιο σχετικά η Συρία πρέπει να το υπογραμμίσουμε είναι μια χώρα στην οποία η θρησκευτική ελευθερία γίνεται σεβαστή έχουμε Ισμαηλίτες, Αλαουίτες, Δρούζους, Χριστιανούς και όλες αυτές οι μειονότητες ε, είναι σεβαστές στην Συρία που είναι μια χώρα πλειοψηφική κασουνιτική και η οποία έχει ένα πολιτικό σύστημα κοσμικού χαρακτήρα και δεν, έχει, δεν προχωράει σε θρησκευτικέ διακρίσεις. Και άμα υπάρχουν εκδηλώσεις ε, ε, κατά της α ή της β κοινότητας τιμωρούνται πολύ αυστηρά. Ενώ σε άλλες χώρες ενθαρρύνονται αυτές οι εκδηλώσεις πολλές φορές και φυσικά δεν τιμωρούνται. Λοιπόν, για τις γυναίκες, η θέση της γυναίκας στο δημόσιο βίο είναι αναγνωρισμένη. Παράδειγμα, η κυρία Ελ Ατάρ είναι η αντιπρόεδρος της Συρίας. Λοιπόν, τώρα, για τους πολίτες των γειτονικών χωρών. Οι σχέσεις της Συρίας με τους γείτονές της έχουν βελτιωθεί σημαντικά. 2008 ε, είχαμε διπλωματικές, τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με το Λίβανο. Και συζητούν οι δύο χώρες μεταξύ τους το θέμα των Λιβανέζων κρατουμένων και αγνοουμένων. Βέβαια τα πράγματα προχωρούν πολύ αργά και αφορούν στην αλλά είχαμε όμως την ανταλλαγή καταλόγων αγνοουμένων όπως επίσης και την απολευθέρωση πολλών κρατουμένων το 2009. Στη Συρία, τώρα με το Ιράκ μιλάμε, στη Συρία έχουμε γύρω στο ένα εκατομμύριο πρόσφυγες από το Ιράκ. Και αυτοί οι πρόσφυγες έχουν όλα τα πλεοκτήματα των πολιτών, των, των υπηκών, σε θέματα δικαιωμάτων, υγείας κλπ και είναι ένα τεράστιο οικονομικό άχθος αυτό για τη Συρία. Τώρα, για τους πολιτικούς αντιπάλους. Η άνοιξη της Δαμασκού δεν ε, απέδωσε τα προσδοκόμενα μακριά από μας. Τα τελευταία χρόνια συνελήφθησαν ε, πολλοί ε, διαφωνούντες, οι κύριοι Σαλέ και Αλμαλέ και όλα αυτά απαγοήτευσαν ιδιαίτερα. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη περιφρούρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συμφωνία Σύνδεσης είναι μια μοναδική ευκαιρία για να συνοδεύσουμε αυτή τη χώρα στην προσπάθεια εξυγχρονισμού πολιτικής και οικονομικής απολευθέρωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας θα εποπτεύει νόμιμα την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία. Ξέρουμε καλά ότι και από την εμπειρία μας με άλλες χώρες ότι το να έχουμε συμφωνία βοηθάει στη βελτίωση αυτών των σχέσεων. Σας ευχαριστώ κυρίως που σεβαστήκατε το χρόνο μιλίας. διότι είχαμε μια καλή συζήτηση για το, με την Προεδρία, αλλά ξεπεράσαμε το χρόνο. Επόμενος προσκεκλημένος, ο κύριος Πόλσον από το Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Euromed. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να σα ευχαριστήσω για το γεγονό ότι μα δώσατε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την παρουσίαση για τη Συρία σε αυτή την υποεπιτροπή. Το δικό μας δίκτυο αποτελείται από 70 οργανώσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στον χώρο της ε, Euromed που δημιουργήθηκε το 1970 σε συνέχεια δηλαδή της συνάψης της μεσογειακής σχέση σχέση στην ε, Βαρκελόνη και ο στόχο προφανώ είναι συνεργασία μεταξύ των ε, ε, διαφορετικών περιοχών και δυνατότητα συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων τη κοινωνίας των πολιτών επιτόπου. Ένας άλλο στόχο μας είναι να ερχόμαστε σε καλύτερη επαφή με τι πρωτοβουλίε και τι διαδικασίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τα ανθρωπίνα δικαιώματα, ούτω ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση σε σχέση με αυτά στις νότιε και ανατολικέ ε, μεσογειακές χώρες. Ε, κατά συνέπεια έχουμε ε, παρακολουθήσει πολύ στενά την κατάσταση στη Συρία κατά τα τελευταία 15 χρόνια και στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, διμερούς συνεργασίας με τη Συρία. Επίσης, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέχισε να εξετάζει την κατάσταση στα ανθρώπινα δικαιώματα στη Συρία και συνέχισε να πιέζει για την απελευθέρωση πολιτικών κρατούμενων στη Συρία με μια σειρά αποψηφίσματα το τελευταίο των οποίων ήταν αφορούσε τον δικηγόρο κύριο Αλ Χασάνη και πέρασε το Δεκέμβριο του 2009. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα την ε, συμφωνία ε, διασύνδεσης με τη Συρία. Τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να προβεί στη σύναψη αυτής της συμφωνίας περίπου πέντε χρόνια μετά από την μονογράφηση αυτής της συμφωνίας. Δυστυχώς η Συρία δεν την έχει προσπογράψει ακόμα, αλλά το γεγονός ότι έχει φτάσει στο σημείο να είναι έτοιμη για υπογραφή μας, δείχνει, μας δίνει, αν θέλετε, μια θετική ε, προοπτική σε ό,τι αφορά δηλαδή και την πρόθεση της εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γνωρίζετε πως εκεί έχει περιληφθεί και το άρθρο 2 το οποίο αναφέρεται ακριβώς στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και θεμελιωδών ελευθεριών καθώς η Συρία έχει κυρώσει όλες τις ε, συμβάσει ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε μια πλατφόρμα για την ε, πολιτική ε, συζήτηση μεταξύ των κυβερνήσεων σε ό,τι αφορά την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς θεωρούμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικυρώσει αυτή τη συμφωνία το ταχύτερο δυνατό γιατί γνωρίζουμε πως αυτό το παράθυρο αν θέλετε αυτή η δυνατότητα ε, συνομιλίας ήταν δύσκολο να φτάσει εδώ που έχει φτάσει. Η κατάσταση σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί μεγάλη πρόκληση ε, στη Συρία. Ε, για να το πω έτσι. Να σας αναφέρω μια σειρά από παραδείγματα. Από το 1963 οι πολίτες της Συρίας ε, ε, ζουν υποκαθεστώς έκτακτο καθεστώς, πράγμα το οποίο βέβαια ε, έχει και πολύ ε, τρομακτικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ελευθερίες. Έχουμε μια, ένα μεγάλο αριθμό από αντιφρονούντες ε, οι οποίοι κρατούνται και έχουμε όχι μόνο τον το δικηγόρο Αλ-Χασάνη αλλά και τον Χάιταμ Αλμάλε ο οποίος ήταν και συνειδητής της νομικού συλλόγου τη Συρία και ο οποίο κρατείται εδώ και κάποια χρόνια. Ταυτόχρονα υπάρχουν απαγορεύσεις μετάβαση ε, στη Συρία και παρακολουθούνται πολύ ε, στενά οι δράσει των διαφόρων ε, επισκεπτών και οι πιέσει αυτέ ασκούνται και στι οικογένειε των πολιτικών αντιφρονούντων. Ε, με βάση τα στοιχεία που έχει το δίκτυό μας ε, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια πρόοδος γιατί καμία οργάνωση από αυτές που τάσσονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχει λάβει επίσημη ε, έγκριση για τη λειτουργία της. Υπάρχουν μας ανεστήρια στις φυλακές, δεν υπάρχει κανένα νέο σε σχέση με χιλιάδες πολίτες οι οποίοι έχουν απλά εξαφανιστεί μέσα στις φυλακές κατά της Συρίας. 300.000 άτομα ε, υπάρχουν τα οποία δεν έχουν επίσημο καθεστώς υπηκότητας, υπάρχουν και μία σειρά ακόμα από τα οποία όμως ε, είμαι σίγουρο πως γνωρίζουν τα μέλη ε, της υποεπιτροπής και μπορούμε προφανώς να σας παράσουμε περισσότερες πληροφορίες αν τις χρειάζεστε. Παρ' όλα αυτά θα θέλαμε να κλείσουμε με ένα θετικό σχόλιο κι εμείς, το ανέφερε ο κ. Μπουρτής, δηλαδή η Συρία έχει επιδείξει μια πιο, πιο θετική στάση έχει αποφασίσει να ε, υποστηρίξει 500.000 ε, ε, Παλαιστινίους αλλά και όλους Ιρακινούς πρόσφυγες. Παρόλα αυτά η κατάσταση σε σχέση με τη Συρία συνεχίζει να ανησυχεί το δίκτυό μας σε αυτό αυτούς τους παράγοντες συγκαταλέγεται το γεγονός ότι δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι στιγμής να δημιουργηθεί ένας διαφανής διάλογος με τις υπηρεσίες της Συρίας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε λοιπόν πως αυτή η εταιρεία συνέσης αποτελεί ακριβώς την ευκαιρία ε, για να υπάρξει ένας τέτοιος ε, ε, διάλογος και θα πρέπει να την πείσουμε πως ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αποτελεί παραβίαση της εθνικής της ασφαλείας και της εθνική τη κυριαρχία. Θεωρούμε πω θα πρέπει να υπάρχει ένα διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Συρία, ο οποίο ε, θα περιλαμβάνει έναν ε, χάρτη πορεία για την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπω αναφέρεται και στο σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Συρία του Δεκεμβρίου του 2009. Ο δικό αυτό χάρτη ε, αναφέρει συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν, για παράδειγμα, άρση τη απαγόρευση μετάβαση από την προσ των ε, όσων τάσσονται υπέρ των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και προφανώς είμαστε στη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε για την περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση τέτοιων στόχων. Θα πρέπει ε, να έρθουμε σε ε, περισσότερη, σε στενότερη επαφή με τη Συρία, ε, διοργανώνοντα συζητήσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υποστηρίζοντα τι οικογένειε των αντιφροντών και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τι δικέ μα κατευθυντήριε γραμμέ σε ό,τι αφορά του όσου προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίση θεωρούμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να υπογραμμίζει τι υποχρεώσει σε ό,τι αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είχε αναλάβει η Συρία στο πλαίσιο αυτή τη συμφωνία σύνδεση. Ε, συνιστούμε το, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξεκινήσει διαλόγους με μέλη του Συριακού Κοινοβουλίου ε, καθώς ε, θεωρούμε πως θα πρέπει να δοθεί συνέχεια σε αυτό το τελευταίο ψήφισμα και στην τύχη του δικηγόρου Αλ Χασάνη και σε τέτοιε συζητήσει προφανώ θα πρέπει να συμμετάσχει και η κυβέρνηση τη Συρία. Τέλο, καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει ένα ψήφισμα υπό τη διαδικασία του καταπίτου, ώστε να ξεκινήσει ένα διάλογο για την έναρξη τη λήψη κάποιων μέτρων για τη βελτίωση της ε, κατάστασης με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, πράγματι, να καλέσουμε εδώ ότι υπήρξε ένα ψήφισμα από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και αναφέρεται και τον κύριο Μουχάναντ Αλχασάνη και να πούμε πως ε, μετά από ένα μήνα είχαμε συναντηθεί με τους ε, εκπροσώπους και με τον δικηγόρο του κύριου Αλχασάνη και γνωρίζουμε πράγματι αυτό που είπατε ότι η Συρία μέχρι στιγμής έχει αρνηθεί να υπογράψει και να κυρώσει τη συμφωνία. τώρα σε ό,τι αφορά τον άλλο ε, δικηγόρο, τον ε, Χαϊτά Μάλε, ο οποίος ε, συνελήφθη στις 14 Οκτωβρίου, έχουμε απευθυνθεί γραπτό στον πρέσβη της Συρίας για να καταδικάσουμε αυτή τη σύλληψη. Ο λόγος τώρα στους συναδέλφους πρώτη έχει το λόγο κυρία Τεκάζα. Δεν ζητήσατε το λόγο. Γιατί είστε πρώτη συγκέντρια για αυτό το ζήτημα. Ε, αυτή η συμφωνία σύνδεσης έχει ε, μαχρόχρονη ιστορία. Περιμένουμε χρόνια αυτή την έκθεση. Εγώ διαδέχθηκα τον Γιάννη ε, Σακελαρίου, ο κύριος Μποντή σε μένα. Και καταφέραμε αυτή, αυτή τη φορά να την πετύχουμε. Άκουσα προσεκτικά την τοποθέτηση του κυρίου Μποντής όπως και τη δική σας και οι δυο έχετε δίκιο στο βαθμό που αν κανείς γνωρίζει καλά την περιοχή αληθεύει ότι μας εκπλήσει η Συρία λόγω ε, ορισμένων ελευθεριών που χτυπούν στο μάτι όμως γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι σκληρό καθεστώς και ότι υπάρχει, γίνονται αυθαίρετες φυλακίσεις πολιτικών αντιπάλων. Μίλησα και τον Μητσελκύλο πριν φυλακιστεί. Εσείς ε, του, του, του, του είχα ρωτήσει εσείς είστε απόλυτα ελεύθερος, είστε εδώ, μου μιλάτε, βέβαια με μικρόφωνα παντού και μου είπε ναι, το καθεστώς μας αφήνει ελεύθερους να κυκλοφορούμε, να μιλάμε για μια συγκεκριμένη φάση, σε μια συγκεκριμένη φάση και μετά στα καλά καθούμε να μας φυλακίζει. Και εμείς περιμέναμε να γίνουν αλλαγές με το συνέδριο του Μπαθ, αλλά δεν έγινε τίποτα για το θέμα της ελευθερίας ε, της έκφρασης. Είχαμε τις ε, δηλώσεις το 2006, τη δήλωση των 300 ε, Συριανών διανομένων που εκφράστηκαν υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης Λοιπόν, ε, ρωτώ, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να συνεργαστούμε με τις αρχές της ε, ε, Συρίας ώστε να βγάλουμε τη Συρία από την απομόνωσή της και από την άλλη να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ συναντήθηκα πολλές φορές με τον Ε, στο, σπίτι του Προέδρου και συζητήσαμε σχετικά ε, προσωπικές υποθέσεις Μερικά άτομα απολευθερώθηκαν μεμονωμένα όμως η συμφωνία θα προχωρήσει πιστεύετε μαζικά τα πράγματα και θα έχουμε ριζικές αλλαγές και να υπάρξει και μια, ε, ένα άνοιγμα του καθεστώτος. και δεν θα ήθελα δεν θα ήθελα εμείς υπάρχει Κατεπίγονα να συνεργαστούμε με, την, ε, με, με, τη Συρία αλλά δεν θα πρέπει να υποσκάψουμε και τις ε, ισορροπίες της περιοχής. Και θα πρέπει να καταλάβει η Συρία ότι πρέπει να αλλάξει πολιτική στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι θα πρέπει να υπάρξουν ανοίγματα. Όπως επίσης ανοίγματα και στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Συμφωνώ με τους δυο σας, γνωρίζω καλά το πρόβλημα και πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε έναν σαφή και ανοιχτό διάλογο. Εμείς είχαμε αυτόν τον διάλογο και στα πιο ψηλά επίπεδα. Ξέρουμε βέβαια ότι είχαμε και τρομοκρατικές ενέργειες, Αλκαΐδα κλπ. Αλλά δεν μπορεί κανείς να, να, μου λέει, όπως μου λέγε τον καιρό εκείνο, ότι ο κύριος Γκίλο ήταν στη ρίζα των τρομοκρατικών πράξεων. Τέλος πάντων ένα μεγάλο πρόβλημα, βέβαια να μην είναι το δέντρο που κρύβει το δάσος. Λοιπόν, ε, ε, υπάρχουν μερικά προβλήματα ελεύθερης έκφρασης, αλλά είναι μια χώρα η οποία είναι αξιοπρόσεκτη στον τομέα των ελευθεριών. Ο κύριος Μπέλντερ, πρόεδρος της αντιπροσωπείας με το Ισραήλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σημερίζομαι την ρεαλιστική αξιολόγηση την οποία έκανε η κυρία Ντοκεζέρ με την οποία είχα τη χαρά να συνταξιδέψω στη Δαμασκό. Ένα ερώτημα προς τους δύο μιλητές μας. Δεν μιλήσατε για τους Κούρδους, αν δεν κάνω λάθος είναι 4 εκατομμύρια. Τι συμβαίνει με τους Κούρδους στη Συρία, τι γίνεται με τα δικαιώματά τους. μιλήσατε για τις θρησκευτικές ελευθερίες. Εγώ σαν χριστιανός, σαν προτεστάντης θα έλεγα ότι η Συρία διακρίνεται με θετικό τρόπο σχετικά με το σεβασμό των θρησκευτικών ελευθεριών. Αυτό ίσως να συνδέεται και με τη φύση του καθεστώτος. Υπάρχει και η εθνική ασφάλεια της Συρίας. Πώς λειτουργεί η υπηρεσία ασφαλείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Διαπιστώνει επίσης κανείς ότι στην ε, Συρία υπάρχουν πάρα πολλοί Ιρακινοί πρόσφυγες οι οποίοι έτυχαν υποδοχής και ανάμεσά τους πάρα πολλοί χριστιανοί. Μιλήσατε για ένα εκατομμύριο. Τα Ηνωμένα Έθνη φτάνουν μέχρι τα δύο εκατομμύρια. Μιλάμε για έναν τεράστιο αριθμό προσφύγων. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικά εξαιρετική επίδοση από πλευράς των Σύρων. Συμφωνώ λοιπόν με την κυρία Ντοκεζέ ότι το πρόβλημα των, του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων παραμένει και ελπίζω εκεί να γίνουν κάποια θετικά βήματα. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει το ρόλο το οποίο καλείται να έχει. Ευχαριστώ κύριε Μπέλντερ. Ο Αντιπρόεδρος έχει το λόγο. Ευχαριστώ και τους δύο μιλητές για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις τους. Και οι παρουσίες του Πάλσεν και οι παρουσίες του Μποντής ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Από ό,τι καταλαβαίνω, και μετά από τα σχόλια τα οποία έγιναν και από την κυρία Κεζεύ μπορούμε να καταλήξουμε εύκολα σε κάποια συμπεράσματα. Η Συρία αντιπροσωπεύει μια πολύ πρωτότυπη κατάσταση θα έλεγα, γιατί από τη μία και πρόσφατα έχει εκδηλώσει την καλή της θα έλεγα πρόθεση για να διαπραγματευτεί μια συμφωνία σύνδεσης και να συνεισφέρει στην ευρωμεσογειακή διαδικασία. Από την άλλη πρόκειται για ένα κράτος το οποίο σίγουρα απαιτείται να κάνει πολλές σημαντικές αλλαγές και σε επίπεδο οικονομικό να περάσει από το σοσιαλισμό στην κοινωνική οικονομία της αγοράς. Το τι θα πετύχει δεν θα το ξέρουμε πριν περάσουν πολλά χρόνια βέβαια. Υπάρχει και το θέμα των προσφύγων, οι οποίοι εμφανίζονται σε μεγάλους ε, αριθμούς θα έλεγα στη Συρία. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιβάρυνση, όπως έλεγε ο Αντιπρόεδρος, ο υπεύθυνο για την οικονομία που ε, μας είχε επισκεφθεί, άκουσα τα σχόλιά του και από ό,τι φαίνεται οι Σύριοι ποτέ δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν ε, στις μεταρρυθμίσεις οι οποίες απαιτούνται αν δεν ξεκινήσουν σωστά ε, για διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων και λόγω της ύπαρξης ενός τόσο μεγάλου αριθμού προσφύγων. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω το εξής ερώτημα στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν ληφθεί υπόψη ε, στα πλαίσια της ε, διαπραγμάτευσης με τη Συρία. Η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καλείται και αυτή να παίξει ένα νέο ρόλο, σημαντικό ρόλο σε σχέση με την ε, υιοθέτηση, μετά από την υιοθέτηση μάλλον της συνθήκης της Λισαβόνας και ακριβώς λόγω του θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εμείς έχουμε πετύχει πάρα πολλές θα έλεγα νέες ε, ε, μορφές αρμοδιοτήτων και συμμετέχουμε στη διαμόρφωση των διεθνών συμφωνιών της Ένωσης. Ευχαριστώ Αντιπρόεδρε γιατί μας θυμήσατε ακριβώς και τον ρόλο τον οποίο και τις αρμοδιότητες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κατά συνέπεια η υποεπιτροπή μας όταν συνάπτονται τέτοιου είδους διεθνείς συμφωνίες. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Και μιας και ο προηγούμενος ομιλητής έθεσε και μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπό της. Α, όχι, έχει ζητήσει το λόγο και η συνάδελφος. Μία ερώτηση για τον κύριο Πάουλσεν. Προφανώς ο διάλογος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά τι σας κάνει να είστε βέβαιος ότι θα πετύχετε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν πολύ σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιστεύετε ότι θα βελτιωθεί η Συριακή κυβέρνηση. Όταν βλέπει άλλους διαλόγους κανείς σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, η κυβέρνηση πολλές φορές για να μειώσει την κριτική ξεκινάει τον διάλογο αλλά μένει στα λόγια, δεν βελτιώνει τα πράγματα. Έχετε θέσει κάποιους στόχους στα πλαίσια του διαλόγου για να μπορέσετε να προσμετρήσετε την επιτυχία του ή όχι. Ευχαριστώ κύριε Λόχπιλε. Πολύ σημαντική η παρατήρησή σας. Γιατί από ό,τι θυμάμαι και η κυρία Ντεκαϊζέρ είχε αναφερθεί στα θέματα στην Τίνιδα. Και εκεί δεν έχουν υπάρξει βελτιώσεις παρά τη συμφωνία. Θα δώσω τώρα λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σχετικά με το πρώτο ερώτημα για το εάν τα συνοδευτικά μέτρα της οικονομικής μετάβασης στη Συρία έχουν ληφθεί υπόψη στη Συμφωνία Σύνδεσης. Ναι, προφανώς. Γιατί η Συμφωνία Σύνδεσης, όπως γνωρίζετε, προβλέπει από τη μία μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συρία και όλες οι, οι ρήτρε τις οποίες έχουμε καταλήξει είναι μεταβατικής ισχύω. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες από πλευρά Συρίας για τη Συμφωνία Σύνδεσης και οικονομικού τύπου. Υπάρχει λοιπόν μία περίοδος μεταβατική η οποία έχει διάρκεια 12 ετή. Υπάρχουν επίσης κάποιες προβλεπόμενες ασυμμετρίες προς όφελος της Συρίας σε σχέση με την τύχη των προϊόντων τους και την εξαγωγή των προϊόντων της Συρίας προς την Ευρώπη. Πρέπει να τα υπενθυμίσουμε όλα αυτά. Υπάρχουν λοιπόν και πάρα πολλά συνοδευτικά μέτρα σε σχέση με την προσαρμογή των δομών της Συριακής οικονομίας. η οποία θα πρέπει να έρθει στο ίδιο επίπεδο αντιμετώπισης των επιχειρήσεων, των κοινωνικών μέτρων γύρω από την αγορά. Όλα αυτά προβλέπονται στα πλαίσια της συμφωνίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σίγουρα να προσφέρει πολλά στα πλαίσια των συναδευτικών μέτρων βοήθειας κάποιων χωρών τόσο συγκεντρωτικών οικονομικά όπως η Συρία προς την ελεύθερη αγορά. Σας έχει τεθεί επίσης και η ερώτηση για τον πολιτικό διάλογο τι εγγυήσεις έχουμε έτσι ώστε ο διάλογος ο οποίος προβλέπεται στα πλαίσια της Συμφωνίας Σύνδεσης να αποδώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα και να βελτιώσει την κατάσταση. Η εμπειρία την οποία έχουμε με τις χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου είναι ότι έχουν υπάρξει βήματα προόδου. Όχι βέβαια στο ύψος των προσδοκιών τις οποίες είχαμε αλλά θα ήθελα μόνο σαν παράδειγμα να αναφερθώ στην περίπτωση της Αιγύπτου όπου πριν από τη Συμφωνία Σύνδεσης και την πολιτική γειτονία και το πρόγραμμα δράσης υπήρχαν λέξεις ταμπού στις συζητήσει μας με τους Αιγυπτίους όπως η διαφθορά, οι συνθήκες κράτησης και όλα αυτά είναι τώρα πλέον θέματα τα οποία συζητάμε ανοιχτά με χώρες σαν την Αίγυπτο γιατί να μην συμβεί κάτι αντίστοιχο και με τους Σύρους. Και εδώ ε, έρχομαι σε αυτά τα οποία είπε στην ανάλυση της η κυρία Ντοκεζέρ. Θεωρούμε ότι οι Σύροι γνωρίζουν τους κανόνες με τους οποίους διαξάγεται ο διάλογος αυτός. Έχουν διαπραγματευτεί λέξη προς λέξη τη συμφωνία αυτή. Η ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αυτή η οποία χρησιμοποιείται συνήθως ο μηχανισμός διακοπής ε, ε, της συμφωνίας αυτής, της ισχύω συμφωνίας αυτής είναι ο προβλεπόμενος. Γνωρίζουμε λοιπόν τους κανόνες, τους γνωρίζουν και οι Σύριοι. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια χώρα με την οποία έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στα πλαίσια του διαλόγου με τη χώρα αυτή. Με τις χώρες γειτονίας βρισκόμαστε πλέον σε αυτό που θα ονόμαζα δεύτερη γενιά των σχεδίων σχέσεων και με τη Συρία δεν έχουμε κάνει υπογράψει ακόμα τη συμφωνία. Υπάρχει λοιπόν ένα πλαίσιο επιφυλάξεων, έλλειψης κατανόησης και ο διόλογος θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια αυτά και να εξηγήσουμε ότι ο διάλογος είναι μια διμερής διαδικασία και θα επιτρέψει να θέσουμε προσυζήτηση και κάποια κοινά σημεία όπως επίσης και σημεία πάνω στα οποία έχουμε διαφωνίες. Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της οικοδόμησης μέτρων εμπιστοσύνης. Και οι επιφυλάξεις και οι καθυστερήσεις οφείλονται ακριβώς σε πάρα πολλά χρόνια έλλειψης επαφών και κατανόησης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποντής έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σημείωσα τις τοποθετήσεις των συναδέλφων. Το θέμα των Κούρδων αναφέρθηκε. Ένα παράδειγμα. Ο μουφτής της Δαμασκού, δηλαδή ο πιο, η πιο σημαντική σουνητική προσωπικότητα της Δαμασκού είναι ένας ε, Σύριος Κούρδος. Το θέμα ότι δεν εξωστρακίζονται οι πολίτες ε, Κούρδοι λόγω της ε, καταγωγής τους. για το δικαίωμα αντιπολίτευσης και ελευθερία έκφρασης. Η εμπόλεμη κατάσταση και το καθεστώς κατοχής ε, στο Γκολάν, η Συριακή επικράτεια, ε, αναφέρεται πάντοτε ως πρόσχημα για κατεξαίρεση μέτρα. Και επειδή φυσικά η σύγκρουση παρατραβάει, ε, γίνεται πλέον κανόνας η εξαίρεση. Εγώ συμμερίζομαι απόλυτα την άποψη της κυρίας Δεκάιζερ, ναι ή όχι συμφωνία σύνδεσης. Η συμφωνία σύνδεσης θα μπορέσει να αποτελέσει ένα διαρκές πλαίσιο συνεργασίας με τους Σύριους, το να απορρίψουμε την ε, συμφωνία, τότε απορρίπτουμε και αυτή με την ευκαιρία για να, για προδεύσει η Συρία. Ευχαριστώ κύριε Μποντής. Ο κύριος Πόλσεν. Ευχαριστώ. Ε, σε ό,τι αφορά ε, το ε, ερώτημα σε σχέση με τους Κούρδους, πράγματι είναι περίπλοκο και υπάρχουν κάποιοι Κούρδοι οι οποίοι πράγματι ε, υπάρχουν μέσα στο, έχουν επίσημα αξιώματα, αλλά υπάρχουν και 300.000 Κούρδοι οι οποίοι δεν έχουν επικοότητα και γνωρίζουμε πως υπάρχει μια νομοθεσία η οποία οθετείται τώρα, ε, η οποία ε, καθιστά αδύνατη ουσιαστικά την αγοραπολισία γης ε, για τους ε, κατοίκους παραμεθόριων περιοχών, πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά την Συμφωνία Σύνδεσης, εμείς δεν είμαστε της άποψης ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει τέτοια συμφωνία. Θεωρούμε ότι είναι σημαντική ε, ε, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, συνεχίσει ε, να, να ασκεί εδώ αυτές τις πιέσεις γιατί ε, με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζει την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακόμα και από δύσκολες συνθήκες. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό όμως να υπάρξουν πλατφόρμες συζήτηση σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί ο μόνος εταίρος αν θέλετε ε, στη Συρία για τις οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οι υπηρεσίες ασφαλείας. Θα πρέπει δηλαδή εδώ να ξεκινήσει ένας διάλογος με πολιτικούς εκπροσώπους της εξουσίας στη Συρία. Ό,τι λοιπόν μπορεί να δημιουργήσει διάλογο σε αυτό το επίπεδο είναι ευπρόσδεκτο. και ίσως μια τέτοια κίνηση ή μια τέτοια προσέγγιση να μην είναι σωστή σε τρία-τέσσερα χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερες πλατφόρμες για διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, νομίζω πως ακούσαμε μια πολύ καλή ανάλυση της κατάστασης και θα πρέπει να δώσουμε μια συνέχεια σε αυτό το ζήτημα και να παρακολουθούμε τις εργασίες ε, εδώ για τις οποίες είναι αρμόδιος ο κύριος Επότη. Ε, και νομίζω πως θα πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε έμβαση και σε αυτό που είπε τώρα ο κύριος είναι δηλαδή ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να θίγουμε πολύ συγκεκριμένε ε, περιπτώσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στα ψηφίσματά μα στι επιστολέ που στέλνουμε στον πρέσβη τη Συρία και ούτω καθεξή. Σα. ευχαριστώ λοιπόν πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στη Συρία πολύ στενά. Ευχαριστώ όλου του συναδέλφου, όλου του ομιλητέ. Τώρα η επίσημη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής τελειώνει εδώ. Θα συνεχίσουμε και κλεισμένο των θυρών χωρίς να πρόκειται για κάτι βέβαια ιδιαίτερα μυστικό αν θέλετε, αλλά θα συνεχίσουμε με τη σύνθεση της υποεπιτροπής ε, που είναι αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τον Εκτρομοκρατισμό και την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρώτη φορά λοιπόν θα έχουμε μια τέτοια συνεδρία με αυτή τη σύνθεση. Πεντάλεπτο λοιπόν διάλειμμα τώρα και μετά μια σχετικά σύντομη συνάντηση αυτής της ομάδας εργασίας. Ευχαριστώ πολύ για αυτήν την συνεδρία. Θεωρώ πως ήταν πολύ καλή αρχή για το νέο έτος.